start with our number 10 of the agenda, that is the civilian CSDP compact, for which I welcome. Ξεκινήσουμε λοιπόν από το σημείο 10, ο Άρνολτ Μόλεναρ, επικεφαλής εμπειρογνώμονας από το CMPD. but I'm sometimes getting at loggerheads with our acronyms. Κάποιες φορές μπερδεύομαι και εγώ με τα ακρόνυμα. Τζοβάνι Φάλεκ, καλώς ήρθατε. Αναλυτής στο EUISS, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για Μελέτες Ασφαλείας. τον πέρατο σε ένα άλλο που ήταν στρατηγικών μελετών και αναπένφρατ εμπειρογνώμας πολιτικής ε, στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διασύνδεσης. με τη συζήτηση που κάναμε για τις ε, αποστολές ΚΕΠΑ τον Ιούνιο, χθε το βράδυ το Συμβούλιο από ό,τι φαίνεται υιοθέτησε ε, το σύμφωνο για αυτές τις επιχειρήσεις πολιτών στο πλαίσιο της ΚΕΠΑ με σκοπό την παροχή ενός νέου ευρωπαϊκού πλαισίου για τη διαχείριση πολιτικών κρίσεων και αποστολών ΚΕΠΑ. Μέσω αυτού του συμφώνου, το Συμβούλιο προτίθεται να αναθεωρήσει τις προτεραιότητες ΦΕΙΡΑ και να τις προσαρμόσει στο σημερινό πλαίσιο και προκλήσεις με τη μετανάστευση, τις υβριδικές απειλές και το καθεξής. Με βάση και τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες EUGS του 2016, το Συμβούλιο θα ενισχύσει το ρόλο του της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ε, φορέα που λειτουργεί με αποτελεσματικότητα και νομιμοποίηση. Πρέπει όμως οι αποστολές πολιτών να ε, αναβαθμιστούν και να γίνουν σύγχρονα και ευέλικτα μέσα εξωτερικής πολιτικής που θα μπορούν να αντιμετωπίζουν ζητήματα ασφαλείας όχι μόνο εκτός Ευρωπαϊκής Υπήρου αλλά και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να το πράξουμε αυτό ε, οι αποστολές ε, πολιτών ΚΕΠΑ θα ε, πρέπει να έχουν και να συνοδευτούν και από μεγάλη προσήλωση και δέσμευση και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, στενότερο συντονισμό μεταξύ κρατών μελών και εξωτερικών φορέων. Επιπλέον, θα πρέπει να ενισχύσουμε και τις ε, αποστολές αυτές και την στήριξη, την ενεργό στήριξη των κρατών μελών. Και από αυτό θα εξαρτηθεί και η επιτυχία τους. Το πολιτικό τμήμα της ΚΕΠΑ είναι πιο περιορισμένο και λιγότερο ορατό από τη θεωρητική διάσταση. Η οθέτηση λοιπόν του συμφώνου ΚΕΠΑ ε, για αυτό το λόγο είναι ένα σημαντικό βήμα προς ε, πιο ε, ευέλικτες και αποτελεσματικές αποστολές πολιτών. Τώρα να δώσω το λόγο στους ε, προσκεκλημένους μας. Να μας πούνε τη δική τους ε, άποψη. Ξέρουμε ότι κάποιες φορές είναι πιο εύκολο να δώσει κανείς διαταγές σε έναν ε, στρατιώτη παρά σε, έναν, ε, σε ένα μέλος του πολιτικού προσωπικού που μπορεί να διαφωνήσει, να φέρει αντιρρήσεις. Φαντάζομαι ότι αν έρχεστε σε επαφή με την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, για παράδειγμα, αλλά όταν υπάρχει πολιτική δέσμευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να δίνουμε και ανθρώπινους πόρους για αυτές τις αποστολές πολιτών. Να δώσουμε πρώτα το λόγο στον κύριο Μόλεναρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που απευθύνατε. για το σύμφωνο αυτό. Όπως είπατε, υιοθετήθηκε χθε από το Συμβούλιο και τα κρατημέλη. Να σταθώ σε αυτό που είπατε στο τέλος. Πράγματι, εντάσσεται σε ευρύτερες προσπάθειες που καταβάλλονται για τη ε, διαμόρφωση μιας στρατηγικής στον τομέα της ε, κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Υπάρχει όμως και μια συμφωνία ορόσημο πλέον ε, για την πλευρά των πολιτών. Εδώ το θέμα είναι ελαφρώς διαφορετικό, γιατί και οι εμπειρογνώμονε που χρησιμοποιούμε για αυτά τα ε, σημεία ε, δεν είναι πάντα, ε, δεν έχουν λάβει πάντα την ίδια κατάρτιση, ούτε είναι πάντα διαθέσιμοι για ανάπτυξη δυνάμεων. Ιδίω στο σημερινό πλαίσιο υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τέτοιους εμπειρογνώμονες σε διάφορα πλαίσια. Εδώ λοιπόν έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό το σύμφωνο είναι το αποτέλεσμα εργασιών που ξεκίνησαν πέρυσι τον Νοέμβριο με πολλά ενδιάμεσα βήματα. Ήδη το Μάιο ξεκίνησε η διαδικασία και είχαμε και το σχέδιο ανάπτυξης ικανοτήτων ε, στις αρχές του εξαμήνου. Το Συμβούλιο έχει τη μορφή συμπερασμάτων του Συμβουλίου και των κρατών μελών πρόσωπα των κατομελών που συναντιούνται ε, στο Συμβούλιο, το οποίο δεν το έχουμε αξιοποιήσει στον τομέα ε, της ε, ΚΕΠΑ, αλλά έχει αξιοποιηθεί σε άλλες, σε άλλες τομείς πολιτικής. Το κάναμε όμω γιατί πολλά από τα ζητήματα που συμπεριλαμβάνονται στο σύμφωνο είναι ζητήματα εθνικής αρμοδιότητας. Γι' αυτό και υπάρχει ρητή αναφορά στα κράτη-μέλη. Αυτά λοιπόν τα κοινά συμπεράσματα δείχνουν τη σημασία του συμφώνου και τη συμμετοχή του Συμβουλίου και των Κρατομελών, φυσικά και τις υπηρεσίες εξωτερικής δράσης και της Κομισιόν. Από πλευράς ουσίας, εμείς εδώ και ένα χρόνο ασχολούμαστε με την προετοιμασία του εγγράφου και όπως είδατε, Έχουμε τρία μέρη σε αυτό το σύμφωνο, στρατηγικές κατευθυντήρες γραμμές. Είναι ένα πολιτικό πλαίσιο δηλαδή. Μετά ένα σύνολο 22 δεσμεύσεων. Και τρίτον, ένα τμήμα που μιλάει για το μέλλον. Για το πολιτικό πλαίσιο και στρατηγικές κατευθυντήρες γραμμές περιλαμβάνει μια σειρά ζητήματα για τα οποία ήδη υπήρχε συνένεση για σύνδεση με την ε, σφαιρική στρατηγική, τις προτεραιότητες για την ενίσχυση ε, της αστυνομίας, του κράτους δικαίου και της διακυβέρνησης σε ε, ασταθείς περιοχές, αλλά και μια ευρύτερη προσέγγιση για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως αναφέρονται και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαΐου. Οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν και κύρια σημεία σε ό,τι έχει να κάνει με τον ρόλο της ΚΕΠΑ σε όλο το κύκλο πολιτικής, τη σημασία της ε, ε τοπικής οικειοποίησης των αποστολών μας, ε, τη σημασία του να έχουμε κλιμάκωση στις επιχειρήσεις, να έχουμε και εκτελεστικές αλλά και μη εκτελεστικές ε, θητείες στις χώρες υποδοχής τη σημασία των μεικτών ε, αποστολών και συνεργασίας μεταξύ στρατιωτικού και μη στρατιωτικού σκέλους και τέλος συνεργασία μεταξύ του τομέα ΚΕΠΑ και δικαιοσύνης και εσωτερικών. Είναι σημαντικό να υπερθυμίσουμε ότι τα ίδια τα καθήκοντα ΚΕΠΑ δεν ε, αλλάζουν. Όμως, ε, ουσιαστικά με το σύμφωνο, θέλουμε να δούμε μήπως μπορούμε να κάνουμε μια καλύτερη και πιο αποτελεσματική ε, χρήση και της πολιτικής αλλά και των ε, καθηκόντων των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από εκείνη. Το σύμφωνο βεβαίως ε, στο επίκεντρό του έχει το σύνολο αυτό των 22 δεσμεύσεων. Όπως είπα, η η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και οι Κομισιόν έχουν αναλάβει το, τα δικά τους καθήκοντα. Έχουμε δομήσει τις 22 δεσμεύσεις με βάση τρεις ε, άξονες, ε, να είναι πιο ικανή η πολιτική, ε, να γίνει καλύτερη χρήση των ικανοτήτων, η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και σε ό,τι φορά την ανάπτυξη ικανοτήτων και την αξιοποίησή τους, μια κοινή προσέγγιση ολοκληρωμένη και συνεργασία με τον τομέα ΔΕΗ. Ο πρώτος άξονας λοιπόν, η πρώτη ομάδα δεσμεύσεων, είναι η πολιτική βούληση και δέσμευση για την ε, οικοδόμηση ε, ικανοτήτων στο πλαίσιο της ΚΕΠΑ. Αυτό είναι ήδη υποχρέωση για τα κράτη-μέλη υπό τη συνθήκη, όπως γνωρίζετε, όμως νομίζω ότι πάντα είναι καλό να το επιβεβαιώνουμε εκ νέου και να διατηρούμε υψηλά το επίπεδο των προσδοκιών παρά και τις εθνικές ανάγκες. Πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των εμπειρογνωμόνων ε, που ε, αποστέλλονται αλλού, γιατί έχουμε δει τελικά ότι ε, έχει περιοριστεί η απόσπαση εμπειρογνωμόνων και χρησιμοποιούνται εξωτερικοί συνεργάτες. Πρέπει να αυξηθεί λοιπόν ο αριθμό ε, των ε, αποσπασμένων. Σημαντική είναι και η βούληση και η δέσμευση των κρατών μελών να δουν τι μπορούν να κάνουν εν είδη βελτίωση στη χώρα του. Και από νομοθετική άποψη και από πλευρά άλλων μέτρων για να μπορούν να διαθέσουν ε, πολιτικούς εμπειρογνώμονες. Και είναι σημαντικό εδώ το Υπουργείο Εξωτερικών να συνεργάζεται με τα Υπουργεία Δικαιοσύνη, Εσωτερικών και άλλα Υπουργεία που μπορούν να παρέχουν εμπειρογνώμονε. Και η κατάρτιση φυσικά είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνη, το οποίο αναδεικνύεται στο σύμφωνο καθώς και η ιδέα ανάπτυξης εθνικών ε, σχεδίων, τα οποία θα ενταχθούν και στην ε, ετήσια διαδικασία αναθεώρησης. Δεύτερος άξονας τώρα για, τις, ε, για την πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των ικανοτήτων μας και να έχουμε πιο καλές αποστολές έτσι. Έχουμε μια σειρά μέτρων με πιο ευέλικτες εντολές. Ένα συλλογικός ποσοτικός δείκτης να έχουμε ε, την ανάπτυξη ε, αποστολής 200 ατόμων εντός 30 ε, ημερών από τη λήψη της απόφασης. Είναι λοιπόν μία εξέλιξη σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ρεαλιστικό στόχος, αλλά αποτελεί και πάλι πρόκληση η ανάπτυξη μιας τέτοιας δύναμης εντός ενός μήνα. Γιατί αυτό προποθέτει και χρηματοδότηση και άλλα πράγματα. Τρίτος άξονας. διασύνδεση αυτών των αποστολών με άλλους ευρωπαϊκούς φορείς, ε, φορείς ε, ΔΕΗ και άλλοι. Είναι σημαντική αυτή η εξέλιξη. Ήδη τα τελευταία χρόνια έχουμε δει βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά πλέον με το σύμφωνο θα το ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο αυτό ούτως ώστε και οι πολιτικέ αποστολέ ε, να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση ε, σοβαρών απειλών και προκλήσεων ή να δίνουν ε, πληροφορίες στις, στους φορείς εθνικής ασφάλειας. Ούτως ώστε να αποβεί αμοιβαία αποφέλη για όλους αυτή τη διαδικασία στα επόμενα χρόνια θα δούμε κατά πόσο μπορούμε να ενισχύσουμε τις ε, πολιτικές αποστολέ αυτή αυτήν την άποψη για να ενισχύσουμε το επιχειρησιακό του αποτέλεσμα. Ίσως δημιουργήσουμε και κάποια πιλωτικά σχέδια στο μέλλον. Όλα αυτά βέβαια πρέπει να τα εξετάσουμε. Μεμονωμένα για κάθε αποστολή και για κάθε χώρα. Τέλος. Το σύμφωνο ε, θέτει και ορισμένες παραμέτρους για την ετήσια διαδικασία αναθεώρησης. Θα τη σχεδιάσουμε βέβαια σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια και το επόμενο συγκεκριμένο βήμα είναι ότι το Συμβούλιο έχει καλέσει την Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερική Δράσης να αναπτύξουν από κοινού ένα σχέδιο δράσης για την υλοποίηση, ε, συνεκτική υλοποίηση του, σχεδίου, του συμφώνου. Μέχρι την άνοιξη του 2019 θα καταρτιστεί αυτό το κοινό σχέδιο δράσης, καθώς και εθνικά σχέδια. Και όλα αυτά θα συμπεριληφθούν ε, στην ε, ετήσια διαδικασία αναθεώρηση. Χθες Υιοθετήθηκε αυτό λοιπόν από τους υπουργούς ε, και αναγνωρίστηκε από όλους ότι είναι μία συμφωνία ορόσημο που δημιουργεί ένα μοναδικό χαρακτηριστικό και λειτουργία της ε, εξωτερικής μας πολιτικής και θα διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό την εξωτερική μας πολιτική για τους επόμενους μήνες και χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε με τον Τζοβάνι Φάλεγκα, ανώτερο αναλυτή Ινστιτούτου Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ασφαλείας. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ την Υποεπιτροπή που με κάλεσε. Συγχαρητήρια σε όλους σας και κυρίως στον κύριο Μόλεναρ για την εκπόνηση αυτού του Συμφώνου Μη Στρατιωτικής Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας. Θα ήθελα να κάνω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις μετά την παρουσίαση του κυρίου Μόλεναρ. Για τα καλά νέα. για το καινούριο βήμα που κάνουμε προς τα εμπρό στη μη στρατιωτική κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, ΚΑΠΑ. Θα ήθελα να σας δώσω κάποια επικοδομητικά στοιχεία για περαιτέρω προβληματισμό και θα ήθελα στο τέλος να δούμε τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε εν ώψη της προθεσμίας του 2023 για την ε, πλήρη υλοποίηση. Να ξεκινήσω λοιπόν με τα πολύ καλά νέα. Έχουμε ένα έγγραφο το οποίο παρουσιάζει σαφή πολιτική στήριξη για μη στρατιωτική κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και για ένα τέτοιο σχετικό σύμφωνο. Πιστεύω ότι είναι ορόσημο αυτό, σημείο καμπής είναι κάτι που χρειαζόμασταν απεγνωσμένα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να γίνει ένα βήμα προς τα εμπρός. Για την πρόληψη των κρίσεων, για τη σταθεροποίηση για τις ε, προτεραιότητες που έχουν ήδη εδρεωθεί σε προηγούμενες σε υψηλό επίπεδο πολιτικές συναντήσεις, για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς έχει αλλάξει ο κόσμος και πώς πρέπει να προσαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την εξωτερική της δράση για να αντιμετωπίσει νέες απειλές. Και όλα αυτά συνάδουν με τους στόχους της συνολική στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την ασφάλεια τη Ένωση, τη ανθεκτικότητα και τη αντοχής των κρατών μελών και των ε, πληγισών περιοχών και τη συμβολή στην Ευρωπαϊκή Ένω... της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση των εξωτερικών συγκρούσεων. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτό εάν δεν έκανε αυτό το βήμα προς τα εμπρός η Ευρωπαϊκή Ένωση, προς την ενίσχυση των, της μη στρατιωτικής κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Και δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίσει τις νέες απειλές, όπως είναι η ριζοσπαστικοποίηση ή ε, το οργανωμένο έγκλημα και οι διάφορες υβριδικές μορφές της τρομοκρατίας έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται στη σημερινή εποχή. Όλα αυτά, λοιπόν, η αποφασιστικότητα αυτή είναι κάτι που πρέπει να μας δίνει ιδιαίτερη ικανοποίηση. Έρχομαι τώρα στις τεχνικές λεπτομέρειες και στην ουσία των δεσμεύσεων. Εδώ, όπως και για οποιαδήποτε πρόοδο και για οποιαδήποτε απόφαση που αποθηκεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ουσία δηλαδή του εγγράφου βασική επίκριση και δεν το λέω για να υποτιμήσω τις προσπάθειες που έχουν γίνει, γιατί πρόκειται για διαπραγμάτευση και μην υποτιμούμε τη δυσκολία στην προσπάθεια εξέβρεση συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Ωστόσο, τα συμπεράσματα είναι πληθωρικά σε λόγια και φτωχά σε αριθμούς. Οι ποσοτικές δεσμεύσεις είναι πολύ μικρότερες. Μπορεί κανείς να περίμενε κάτι διαφορετικό. Κατά πάσα πιθανότητα όχι. δεν θα μπορούσε να περιμένει τα συμπεράσματα να είναι πολύ συγκεκριμένα από πλευράς δεσμεύσεων. Παρ' όλα αυτά, έχουμε κάποιες ενδείξεις για το ότι πέραν όλων αυτών που έχουν δηλωθεί και έχουν τύχει στήριξη από τον πολιτικό λόγο, τον δημόσιο, τώρα θα έλθει η φάση της υλοποίησης. Τι θα κάνουμε δηλαδή με αυτές τις πολιτικές δηλώσεις. Δεν θέλω να υποτιμήσω το γεγονός ότι ε, κάτι που είναι σημαντικό είναι η πολιτική διακήρυξη, οι πολιτικές δηλώσεις. Αυτό είναι σημαντικά. Έχει έρθει ώρα όμως να μπούμε στην ουσία, στον πυρήνα του θέματος, να δεσμευτούν τα κράτη-μέλη. Να υλοποιήσουν τις υποσχέσεις που έχουν δώσει και τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει. Εδώ λοιπόν τα νέα είναι λιγότερο ίσως ευβίωνα. Δεν είναι κακά βέβαια. Έχουμε το ποσοστό των εθνικών εμπειρογνωμόνων που αυξάνεται. Δεν λέω ότι αυξάνεται ριζοσπαστικά, αλλά εν πάση περιπτώσει δημιουργεί ένα σημείο αναφοράς. Έτσι θα έχουμε εθνική εμπειρογνωμοσύνη στις μη στρατιωτικέ αποστολέ κοινή πολιτική ασφάλεια και Άμυνα. Και παρόλο που δεν υπάρχει συγκεκριμένο νούμερο για το πόσα έτη συγκεκριμένα σε πόσα έτη θα εκτυλιχθεί όλο αυτό το πρόγραμμα, έχουμε μεγαλύτερη ανταπόκριση και μεγαλύτερη ευελιξία εάν εφαρμοστούν σωστά οι συστάσεις που περιλαμβάνει το σύμφωνο αυτό. Επίσης θετικό είναι το γεγονός ότι δίνεται όθηση σε περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων που έχουν να κάνουν με τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων για θέματα και εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Και αυτό είναι θεμελιώδες όχι μόνο από την τεχνική σκοπιά του θέματος, αλλά και για τις πολιτικές προεκτάσεις που θα έχει αυτή η δράση. Γιατί επανειλημμένως έχω πει ότι το, το σύμφωνο μη στρατιωτική κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα και όχι εξωτερική, δεν πρέπει να περιοριστεί στη μετανάστευση και σε αυτό το φαινόμενο μόνο, αλλά ε, θα πρέπει να επεκταθεί και να βγάλει ρίζες, να ριζώσει. Γιατί είναι βασική λογική, ε, αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό στοιχείο του δημόσιου πολιτικού λόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι μπορούμε να περιμένουμε τους επόμενους μήνες και χρόνια τώρα. Το έγγραφο το δηλώνει ξεκάθαρα. Κοινή δράση, κοινό σχέδιο δράσης μέχρι την άνοιξη του 19 από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά, εθνικά εφαρμοστικά σχέδια που θα ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένη μορφή που θα διαμορφωθεί το, σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Ε, ε, ενδιάμεσες αναθεωρήσεις αιτήσιες από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για να έχουμε κίνητρα αλλά και δείκτες για τη μέτρηση των επιδόσεων των κρατών μελών και για να ξέρουμε κατά πόσο τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν τις συστάσεις του συμφώνου και ενδιάμεση αναθεώρηση για να αποτιμηθεί η πρόοδος που θα έχει σημειωθεί. Τα βασικά και τα γνωστά δηλαδή, τα κλασικά πέρα από τα εθνικά εφαρμοστικά σχέδια, ποιο θα ήταν το κίνητρο για τα κρατη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Και αν τελικά δεν ε, φέρουν αποτελέσματα και αν πούν τα κράτη-μέλη ναι στα λόγια και στην πραγματικότητα δεν γίνει τίποτα. Και αν τελικά έρθουν τα κράτη-μέλη και πούν όχι. Δεν είδα ενδείξεις για τον προϋπολογισμό. Δεν υπάρχει σαφής δέσμευση να αυξηθεί ο προϋπολογισμός. Ίσως αυτό θα ήταν πολύ υπερβολικό να το περιμένουμε από ένα τέτοιο είδους έγγραφο. Ωστόσο, αν θέλουμε να έχουμε σοβαρές φιλοδοξίες, τότε το λανθάνον ερώτημα είναι πώς χρηματοδοτούνται οι φιλοδοξίες. Ε, αυτό το ερώτημα κάποια στιγμή πρέπει να απαντηθεί και να δοθούν νέα μέσα και να επιδείξουμε και μια κάποια δημιουργικότητα, γιατί όχι. Τώρα, γενικά ως προς την ευελιξία και την ευθυγράμμιση στη διαδικασία ε, λήψης πολιτικών αποφάσεων, όλα αυτά είναι σημαντικά και πρέπει να δούμε πώς θα επιτευχθούν. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί. Με ποιους μηχανισμούς μπορεί να υπάρξει περισσότερη ευελιξία στην μελλοντική κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Τελικά, αυτό που θα έπρεπε να περιμένουμε, εκτός από αυτό που μπορούμε να περιμένουμε τους επόμενους μήνες, είναι το εξής. Τα κράτη-μέλη θα τηρήσουν αυτή την πολιτική συνένεση για τη μη στρατιωτική κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ναι, θα επιταχύνει, θα εντείνει τις προσπάθειές της και θα δράσει ως ένας θαυμάσιος διαμεσολαβητής και θα ασκήσει πίεση στα κράτη-μέλη για να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και θα γίνουν και πιο συγκεκριμένες συζητήσεις για το οικονομικό σκέλος. Αυτό, αυτά είναι τα σίγουρα δηλαδή. Και όσοι δεν διάβασατε την ενημέρωση της Νικολέτα Πυρότση που είναι στην ιστοσελίδα τη σχετική για το Σύμφωνο Μη Στρατιωτική Κοινή Πολιτική Ασφάλεια και Άμυνα, εκεί όπου χαρακτηρίζεται δηλαδή αυτό το σύμφωνο ω μια ιστορία επιτυχία, επιτρέψτε μου να σας αναφέρω τα συμπεράσματά της και παραθέτω τα λόγια σας, τα λόγια της. Πιστεύω ότι η συζήτηση και η διαδικασία που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο, πράγματι έδωσε το γενικότερο πλαίσιο σε αυτή την πολιτική ασφάλειας και άμυνα, το ενιολογικό πλαίσιο για να αναπτυχθεί αυτή η δράση και πράγματι έδωσε σε αυτή την πολιτική τις νέες δυνατότητες, το ενδεχόμενο δηλαδή να αξιοποιηθούν, να διερευνηθούν, να βελτιωθούν οι δράσεις και οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνονται σε αυτό το πλαίσιο και αυτό το έγγραφο έρχεται τώρα για να δώσει μια συλλογική πολιτική δέσμευση και στήριξη. Σε αυτό χρησιμεύει αυτό το έγγραφο. Αυτό το οποίο όμως που δεν έχουμε και που θα πρέπει να παρακολουθούμε προσεκτικά είναι η διασφάλιση, η διαβεβαίωση ότι αυτές οι δεσμεύσεις θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και αυτό το οποίο αναγράφεται επί χάρτου σήμερα εδώ μέσα σε αυτό το έγγραφο θα εφαρμόζεται και θα έχουμε σωστά ε, αντισταθμιστικά στοιχεία ελέγχου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα θεσμικό όργανο που μπορεί να αναλάβει πιο δραστήριο ρόλο στο τομέα της ασφάλειας, της άμυνας, αλλά και στο μη στρατιωτικό σκέλος της ασφάλειας. Και πρέπει η εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να είναι πιο σημαντική, να πλησιάσει σε αυτή τη διαδικασία, να έχει σωστή τροφοδότηση, σωστή παρακολούθηση και συμβουλευτική, να διασφαλίσει δηλαδή το Κοινοβούλιο ότι η διαδικασία που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο ολοκληρωθεί, ε, ότι θα ολοκληρωθεί με επιτυχία μέχρι το 2023 για να μπορέσουν οι προσδοκίες μας από αυτό το σύμφωνο να αποδειχθούν αληθινές. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται να μας καλέσετε δύο φορές και με την πρώτη αυτή πρόσκληση θα ανταποκριθούμε. Η κάθε φορά που χρειάζεται κάτι να ελεγχθεί, είμαστε εμείς εδώ ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θεωρούμε ότι είναι ένα από τα καθήκοντά μας να ε, το παρακολουθούμε στενά. Ευχαριστώ. Έρχομαι τώρα στην κυρία Άννα Πένφρατ υπεύθυνη πολιτικής. Εγώ εργάζομαι για την ΕΠΛΟ, ε, που είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Σύνδεσμος για την Οικοδόμηση της Ειρήνης. Ε, και ο στόχος μας είναι να προλάβουμε βίες ε, συγκρούσεις. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να πω μερικά λόγια σχετικά με το σύμφωνο αυτό και κυρίως με τη διαδικασία που οδήγησε στο σύμφωνο. Και μετά θα σας παρουσιάσω βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη αν επιτιμούμε οι αποστολές να είναι επιτυχημένες, να συμβάλλουν στη βιώσιμη ειρήνη και επίσης το τι είναι απαραίτητο να γίνει κατά την εφαρμογή και τι πρέπει ακριβώς να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, θα ήθελα να υπογραμμίσω κυρίως κάποιες έννοιες όπως πάμε το χάρη ε, το να προαγεί κανείς την οικειοποίηση του προγράμματος ή την ε, ασφάλεια των ανθρώπων. Ξεκινάω λοιπόν με το σύμφωνο και τη διαδικασία που οδήγησε σε αυτό. Υπάρχουν ε, κάποιες ανησυχίες πριν εφαρμοστεί το σύμφωνο σχετικά με την ισορροπία που πρέπει να επικρατεί αφενός όσον αφορά την εσωτερική ασφάλεια, αυτό που πιστεύει κανείς γι' αυτό, και από την άλλη με την πρόκληση ασφάλειας που αφορά όλους τους πολίτες, ε, θέματα όπως η τρομοκρατία, η μετανάστευση. Δεν είναι απαραίτητα θέματα ασφάλειας ή θέματα προτεραιότητα. Ε, αυτό το έδειξαν βέβαια και άλλοι ομιλητές, αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά από το να κάνει κανείς ε, το σύνδεσμο ανάμεσα στην εσωτερική ασφάλεια σε πολιτικό επίπεδο και να μεταφέρει όλη τη raison d'être των αποστολών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί μακροπρόθεσμα αλλά και μεσοπρόθεσμα να βλάψει τη δική της την ασφάλεια αν εστιάσει σε βραχυπρόθεσμα ωφέλη από το θέμα της μετανάστευσης. Νομίζω αυτά έχουν συζητηθεί ευρέω, γιατί υπάρχουν τομείς ε, όπου τέτοιου είδους θέματα αποτέλεσαν boomerang, παραδείγματος χάρη μελέτες που υπάρχουν σήμερα σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις ε, της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ιγυρία ή ε, επίσης ε, το ε, πώς τέτοιου είδους αντιδράσεις μπορούν να οδηγήσουν σε αντίμετρα. Νομίζω ότι όλα αυτά οδήγησαν σε πολλές συζητήσεις και θα ήθελα να πω ότι τελικά οι στρατηγικές κατευθυντίες γραμμές είναι αρκετά ισορροπημένες. Με την έννοια ότι τονίζουν τις προτεραιότητες, και επίσης ε, θα ήθελα να φέρω και τη σημασία του το πόσο έχει σημασία να οικειοποιηθεί κανείς ε, αυτό το πρόγραμμα η προκαταρκτική διαδικασία μπορεί και αυτή να οδηγήσει στο να μείνουν κάποια ίχνη. Άκουσα ότι έγινε λόγος ε, για την ε, μη στρατιωτική πολιτική ασφάλειας και άμυνας ε, σχετικά με την ιεράρχηση στην οποία προβαίνει εκείνη και θέλω να σας πω ότι ήδη υπάρχει διαφορετική ερμηνεία των αποστολών. Διαφορετικά ο καθένας ερμηνεύει μια αποστολή. Εάν λοιπόν αυτή η έννοια της, ε, του σχεδιασμού της MBTP ε, εφαρμόζεται. Νομίζω ότι ένα βασικό στοιχείο είναι να ξεκαθαρίσουμε ότι οι αποστολές ε, της ασφάλειας και της άμυνας έχουν ως στόχο την ασφάλεια των πολιτών. Και εδώ εννοούμε ότι το θέμα δεν είναι να ενισχυθεί το κράτος ή οι τοπικές δυνάμεις, αλλά αυτό που παίζει ρόλο είναι να αντιμετωπιστούν οι διάφορες προκλήσεις που μπορούν να αφορούν ε, τις ε, ε, φιλοξενούσες χώρες. Η έννοια της ανθρώπινης ασφάλειας δεν υπάρχει στο σύμφωνο και δυστυχώς αυτό οφείλεται στο ότι βεβαίως και αναφέρεται η παγκόσμια στρατηγική ή ε, τα έγγραφα για την εφαρμογή αυτής της ε, πολιτικής. Όμως ε, αναφέρεται και η ανθρώπινη ασφάλεια για να διευκρινιστεί τι είδους ασφάλεια και σταθερότητα ε, προσπαθεί να προάγει αυτή η μη στρατιωτική πολιτική ασφάλειας. Νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει είναι να προχωρήσει αυτή η όλη συζήτηση για την πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι τα βασικά στοιχεία έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικές οι πολιτικές ε, και σε ποιο βαθμό εξετάζονται όλα αυτά στο σύμφωνο. Να λοιπόν ότι εδώ δεν λέω ότι η πολιτική αυτή θα πρέπει να είναι ένα μακροχρόνιο εργαλείο, αλλά να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το εργαλείο διαχείρισης κρίσεων μπορεί να συμβάλλει στην δρέωση της ειρήνης. Και είναι σημαντικό να επενθυμίσουμε σε όλους ότι οι αποστολές της πολιτικής αυτής πρέπει να έχουν ένα θετικό αντίκτυπο. Γιατί πολλές φορές τις συζητήσεις βασίζονται στην παραδοχή ότι οι παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξορισμού είναι θετικές. Όμως, ε, ακόμα και ο καλύτερος σχεδιασμός επί χάρτου, ε, ακόμα και αν γίνεται στις Βρυξέλλες, μπορεί να αποτύχει εάν το περιβάλλον είναι τροτό και βάλιτο, όπως αυτό μέσα στο οποίο αναπτύσσονται αυτές οι επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν που ενδιαφέρει είναι από το να σε επίπεδο αποστολής και να αντιμετωπίσετε καλύτερα το περίπλοκο του περιβάλλοντος, αλλά όπως επίσης ε, και οι ε, συνέπειες των δραστηριοτήτων και εσκεμμένες συνέπειες. Άρα δηλαδή πρέπει να προάγουμε στοιχεία που έχουν ήδη αναφερθεί προηγουμένω, μεταξύ αυτών η ανθρώπινη ασφάλεια που μπορεί να σας φέρονται αυτονόητα, αλλά αν μιλήσετε με διάφορους ανθρώπους που μιλάνε για την πολιτική αυτή, ε, θα ακούσετε και πάρα πολλές και διαφορετικές έννοιες για το τι σημαίνουν αυτοί οι ορισμοί, αυτά τα στοιχεία. Εμείς ε, έχουμε επενδύσει και σε κάτι άλλο, στην αποκαλούμενη ευαισθητοποίηση για τις ε, συγκρούσεις. Νομίζω αυτό αναφέρεται και στην ε, παγκόσμια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού που νομίζω ε, δεν είσαστε όλοι εξοικειωμένοι, γι' αυτό πρέπει να ε, τα εξηγήσουμε λίγο. Η ευαισθητοποίηση σημαίνει ότι επενδύουμε σε μια ενδελεχή ανάλυση του πλαισίου μέσα στο οποίο αναπτύσσεται μια προστολή. Ε, η ανάλυση αυτή συνεχίζει και κατά τη φάση της εφαρμογής. Το δεύτερο στοιχείο είναι να υπάρχει επαρκής έλεγχος και μηχανισμός αξιολόγησης έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής αξιολόγηση των επιπτώσεων μιας αποστολής στη δυναμική των συγκρούσεων για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα προκύπτει ζημιά και θα μαγιστοποιούμε το κέρδος. Το τρίτο είναι να υπάρχει η δυνατόν προσαρμογή των ε, εξελίξεων της χαρασόμενης πολιτικής. Ε, έλεγχος και προσαρμοστικότητα, ε, η ανάλυση βεβαίως και παίζει ρόλο για θέματα συνδυτοποίησης και αυτό νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο. Βέβαια, οι επενδύσεις στην ανάλυση μπορούν ε, να βελτιωθούν κατά την εφαρμογή, αλλά αυτό πρέπει να το δούμε στη φάση του σχεδιασμού. Επίσης, αυτό που ενδιαφέρει είναι πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε όλες οι προοπτικές και αυτές τις ε, κοινωνίες των πολιτών ε, μπορούν να συμπεριληφθούν. Όσον αφορά τον έλεγχο και την αξιολόγηση, υπάρχει ένα στοιχείο, το στοιχείο υπαριθμών 13 στο σύμφωνο, που ε, περιλαμβάνει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Βεβαίως θα πρέπει να δούμε τη σημασία που θα αποδοθεί στα διάφορα προγράμματα εφαρμογής. Γιατί πρέπει να ομολογήσω ότι ότι ε, δεν είναι εύκολο να εφαρμόσει κανείς ε, ένα πρόγραμμα δράσης σε ευρύτερη κλίμακα. Ούτε είναι εύκολο να υπάρχει σωστή αναφορά κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Άρα δηλαδή επ' αυτού πρέπει να υπάρξουν Το τελευταίο είναι η προσαρμοστικότητα, το ανέφερε ο Τζοβάνι και ο Άρνολτ. Υπάρχουν πολλά στοιχεία στο σύμφωνο για την προσαρμοστικότητα, την ευελιξία, την κλιμάκωση. Αυτά είναι πολύ σημαντικά εργαλεία που πρέπει να δοκιμαστούν. Και θα δούμε σε ποιο βαθμό οι επιχειρήσεις μπορούν και αυτές να προσαρμοστούν μετά από την αξιολόγηση και τον έλεγχο ε, αντί να δίδονται, αποδίδονται πολιτικά στοιχεία σε αυτό το εργαλείο, σε αυτό το μηχανισμό. Να ανακεφαλαιώσω λιγάκι τι σημαίνουν όλα αυτά για τα εθνικά προγράμματα και για την ε, ε, τήσια ε, αναθεώρηση. Το ένα είναι η γλώσσα, δηλαδή να υπάρχει η έννοια της ανθρώπινης ασφάλειας, να συμπεριλαμβάνεται αυτή η έννοια. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό. Όσον αφορά τις ικανότητες, αναφέρομαι στο 70% που αναφέρθηκε και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να οικειοποιούνται τα προγράμματα. Η τεχνογνωσία και η ανάλυση των συγκρούσεων, ε, τα δικαιώματα, ε, η αναγνώριση και η ισοτιμία των δύο φύλων. Αυτά όλα είναι προσδοκίες για τα οποία ε, μερικές φορές είναι δύσκολο να συμπεριληφθούν στην πολιτική της, ας πούμε, του Υπουργείου Εσωτερικών ή του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Είναι λοιπόν να διασφαλιστεί ότι αν τελικά θέλουμε να επιτύχουμε αυτό το στόχο του 70%, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βουτάνε, επιτρέψτε μου την έκφραση, ε, σε άλλα αποθεματικά από ότι ορισμένα υπουργεία, ε, τα οποία οποία έχουν και αυτά βέβαια κάποια τεχνογνωσία ε, γιατί έχουν εκπροσώπους τους ε, στα, ε, στην κοινωνία των πολιτών ή οπουδήποτε αλλού. Κάτι άλλο. Πρέπει να υπάρχει και χώρος κατά την εφαρμογή, έτσι ώστε να συζητούνται κυρίως οι βέλτιες πρακτικές για τον έλεγχο, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των επιπτώσεων. Και ξέρω ότι γίνονται πολλές συζητήσεις για την εκπαίδευση, αλλά πέρα από την προαγωγή της παραδοσιακής εκπαίδευσης, ε, μπορούμε να αναφερθούμε και σε προγράμματα τα οποία μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμα και αφορούν το προσωπικό. Και θα τελειώσω αναφερόμενοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να βοηθήσει με πάλους τρόπους. Ε, πρώτον, να έχει μια συζήτηση έτσι ώστε να προάγει τι έννοιες ε, τη ανθρώπινη ασφάλειας μεταξύ άλλων. Δεύτερον, να διασφαλιστεί η πολιτική πίεση σε ενωσιακούς θεσμούς για να γίνονται αναλύσεις, να υπάρχει έλεγχος, να εξάγονται συμπεράσματα, να, ε, να εντοπίζονται οι βέλτιστες ε, πρακτικές. Σημασία έχει να διασφαλίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι θα εξάγει συμπεράσματα με αυτά, σε σχέση με αυτά τα οποία βιώνει. Και κάτι άλλο, όταν υπάρχουν ακροάσεις με τους επικεφαλείς των επιχειρήσεων ή και με άλλους εμπειρογνώμονες, να μπορεί κανείς ε, να ε, υποβάλει συγκεκριμένες ερωτήσεις για συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Και νομίζω ότι αυτό εδώ έχει σημασία να συμμετέχουν και άλλοι εξωτερικοί, ε, εξωτερικοί εμπειρογνώμονες. Μιλάει πάρα πολύ γρήγορα η μιλήτρια, πράγματι. Έτσι λοιπόν να υπάρχουν ε, συναντεύξεις ε, και συζητήσεις ε, με επικεφαλής των επιχειρήσεων για να μπορεί να γίνει μια αξιολόγηση. Σας είπα ότι είναι σημαντικό σε αυτές τις συζητήσεις να συμμετέχουν και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες. Και τέλος, ίσως θα πρέπει κανείς να βουλέψει πάνω στο πώς μπορεί να οργανωθεί καλύτερα μια επιχείρηση. Εδώ μπορεί να συνεργαστεί με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, παραδείγματος χάρη. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω επανερχόμενοι στο γιατί είναι σημαντικό να επενδύει κανείς στην ασφάλεια, τη τοπική κοινωνία στις χώρε με τι οποίε συνεργαζόμαστε και να μεριμνούμε έτσι ώστε να ε, λειτουργούμε σωστά με την απαραίτητη ευαισθησία. Αυτό είναι σημαντικό γιατί βεβαίω και είναι κανονιστική αν θέλετε δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αν δείτε λιγάκι όλε τι συνθήκε, αλλά και διότι με τον τρόπο αυτό οι δράσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται πιο αποτελεσματικέ και έτσι μπορεί κανεί να συμβάλλει σε μια βιώσιμη ειρήνη για όλου του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποιοι λείπουν, η συνάδελφος Βαλέρη όμως είναι εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για τις ε, παρουσιάσεις σας. Είμαι θετικά διακείμενη ε, προ μια μεγαλύτερη εστίαση προ αυτέ τι αποστολέ. Είναι κάτι το οποίο έχουμε ζητήσει εδώ και πολύ καιρό. Ελπίζω να συνοδευτεί και από τον κατάλληλο προπολογισμό όταν φτάσουμε εκεί. Έχω όμω ορισμένα ερωτήματα. Πρώτον, για τη μεγαλύτερη ικανότητα σε ό,τι αφορά το μη στρατιωτικό σκέλο. Ε, είπαμε ότι χρειαζόμαστε πολύ κατάρτιση, στήριξη και το καθεξής αυτή τη στιγμή, σε αυτή την περίπτωση, βασιζόμαστε περισσότερο στην, ε, στο κράτος δικαίου. Χρειαζόμαστε αστυνομία, δικαστές και ξέρουμε ότι έχουμε ελλείψεις στη δυνατότητα κατάρτισης και βούλησης κάποιες φορές από τα κράτη-μέλη να τους αφήσουν. Είναι σημαντικό λοιπόν να το εξασφαλίσουμε αυτό. Μίλησα με αστυνομικού στη Σουηδία πριν από πολλά χρόνια, γιατί υπήρχε τότε το ζήτημα αν θα πάμε στο Αφγανιστάν να ε, εκπαιδεύσουμε την αστυνομία. Μας είπαν ότι είναι επικίνδυνο, ότι είχαν πολλά προβλήματα με τις ε, άδειε από την Σουηδική αστυνομία, γιατί και εμείς έχουμε έλλειψη αστυνομικών και δεν το βλέπουν σαν κάποιο προσόν την αποστολή που έχουν κάνει για ένα εξάμεινο. Πρέπει λοιπόν ε, να κάνουμε πολλή δουλειά εδώ. Για το δικαστικό σκέλος είναι ακόμα πιο δύσκολο ίσως να τους πείσουμε να πάνε. Αύξηση της, ε, του feedback, της ανατροφοδότησης για πολλές χώρες, όπως και στο Αφγανιστάν. Ζητήσαμε μήπως μπορούσαμε να πάρουμε αστυνομικού από το Αφγανιστάν και να του φέρνουμε στη Σουηδία για να του εκπαιδεύσουμε. Ίσως ήταν πιο εύκολο έτσι. Αυτή ήταν μια ιδέα που είχε ε, ακουστεί τότε. Είναι σημαντικό να το λύσουμε αυτό. Τώρα για... Κοινέ προσπάθειες και συνεργασία. Μιλήστε για συνεργασία με ε, τον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Μιλήστε για τη μετανάστευση. Τα πρώτα σημεία εδώ είναι ότι πρέπει να ζητήσουμε από την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσουν ένα σχέδιο δράσης. Γιατί τα περισσότερα σχέδια δράσης αυτή τη στιγμή που επικεντρώνονται στην ε, ε, αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Αυτό βλέπουμε και εδώ στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Πολύ φοβάμαι λοιπόν ότι όλη αυτή η προσπάθεια θα εξαντληθεί εκεί, στα σύνορα. Θέλω να μας πείτε κάτι παραπάνω. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση Γιατί κατά τη γνώμη μας, όταν φτάνουν οι μετανάστες ε, στις ακτές της Μεσογείου ή ακόμα και στα σύνορα ε, Λιβύης, Νιγηρά, φτάνουν εκεί επειδή... Νιγηρίας, ε, τότε το πρόβλημα έχουμε ήδη αποτύχει, γιατί σημαίνει ότι δεν έχουμε κάνει αρκετά για να αποτρέψουμε ε, και να διορθώσουμε τις συνθήκες που τους εξωθούν σε αυτές τις κινήσεις. Δεν λύνονται δηλαδή αυτά τα προβλήματα στα σύνορα. Και γι' αυτό βλέπω ότι έχουμε πολλά ε, project στα σύνορα και αυτό μας στερεί πόρους από αλλού. Επομένω, ελπίζω να μας πείτε κάτι παραπάνω για τη συνεργασία ε, στον τομέα ΔΕΗ. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος να πάρει το λόγο. Εάν όχι, να προστάσω κι εγώ κάτι. Πραγματικά δεν ρωτώ με ποιο είναι το καινούριο στοιχείο σε σχέση με τους στόχους που είχαμε από το 2000. Αλλά και πέρσι στην ετήσια έκθεση διαπιστώσαμε με, με τα ότι δεν έχουμε επαρκές πολιτικό προσωπικό που να παρέχεται τα κράτη-μέλη και αυτός ο στόχος ακόμα δεν έχει επιτευχθεί. Επομένως, δεν έχουμε πετύχει καν τους παλιούς στόχους. Τώρα ορίζουμε νέους. Γιατί να θεωρήσουμε ότι τώρα το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη θα πετύχουν ε, τους στόχους και θα εκπληρώσουν τα υπεσχημένα. Αφού δεν το έχουν πράξει μέχρι τώρα. Εάν όντως έχουν σοβαρό σκοπό εδώ τα κρατη Αυτό θα πρέπει να αντικατοπτριστεί και στη συζήτηση για τον προπολογισμό του 2019. Εκεί είναι πραγματικά η απόδειξη ότι έχουν πάρει στα σοβαρά αυτή την υπόθεση. Αν λοιπόν ε, τα αντιμετωπίζουμε σοβαρότητα, πρέπει να βρουν και τους απαραίτητους πόρους. Η τελευταία έκθεση από το ελεγκτικό συνέδριο μας έδειξε τους περιορισμούς ε, αυτών των αποστολών. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει πρόβλημα σε τρίτες χώρες. ως προς τον αντίκτυπο στους ε, αρμόδιους ε, πολιτικούς θεσμούς. Ξέρετε ότι αυτό, νομίζετε μάλλον ότι αυτό θα αλλάξει με αυτό το σύμφωνο. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο. Ωραία. Ο κύριος να και πάλι. Ευχαριστώ. Φυσικά και το σύμφωνο είναι μια συμφωνία ορόσημο, αλλά δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα αποτελέσει πανάκια για όλα τα προβλήματα. Είναι μόλις η αρχή, λοιπόν. Τα θέματα που θίξατε είναι θέματα που έχουμε συζητήσει και μεταξύ κρατών μελών. Και εδώ προσπαθούμε να βρούμε την ισορροπία μεταξύ μια ε, κλασικής προσέγγιση σε αυτά τα ζητήματα και σε ποιο βαθμό μπορούμε να εξετάσουμε αυτές τις ενέργειες στο πλαίσιο και των αναδυόμενων προκλήσεων και κινδύνων και πού ακριβώς ε, βρίσκουμε αυτή την ισορροπία ή αποστολές ε, και ΕΠΑ. Έχουμε κάνει πολλά πράγματα ήδη τις τελευταίες δεκαετίες σε αυτόν τον τομέα. Προσπαθούμε λοιπόν να ξεφύγουμε από ε, αυτή την αντίφαση μεταξύ νέου και παλιού. Παράλληλα, προσπαθούμε να δούμε κατά πόσο οι ενέργειες αυτές θα είναι προς το, συμφέρον μας ή προς το συμφέρον ε, του τοπικού πληθυσμού, της τοπικής κυβέρνησης και του καθεξής. Το ιδανικό θα ήταν να είναι αμοιβαία αποφελής. Και λέμε ότι με την ε, προώθηση της ασφάλειας επιτόπου αυτό έχει αντίκτυπο και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Τώρα όμως, όταν ε, εξετάζουμε το θέμα με τα Υπουργεία στην τομέα ΔΕΗ που πρέπει να αποσπάσουν το δυναμικό τους και να το στείλουν εκεί. Ε, εκεί διαφέρει το πράγμα. Υπάρχει λοιπόν όλη αυτή η συζήτηση. Τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω. Για, από, για να δώσουμε κίνητρα στα Υπουργεία να αποστείλουν προσωπικό παρά τις εθνικές τους ε, ανάγκες. Επομένω, στο μέλλον θα πρέπει να σταθούμε σε, αυτές τις, σε αυτά τα κίνητρα και πολιτικά αλλά και οικονομικά. Δεν είναι απλό γιατί ο προπολογισμό εντάσσεται στην εξωτερική δράση. Δεν μπορούμε λοιπόν με αυτόν τον προπολογισμό να βοηθήσουμε την ανάπτυξη ικανοτήτων ε, στα κρατη Πρέπει να δούμε αν μπορεί να υπάρξει συνέργεια με τον κλάδο ΔΕΗ για να καταρτήσουμε συνοριοφύλακες και το καθεξής. Μπορούμε να βρούμε λοιπόν κάποιον τρόπο για να τους βοηθήσουμε. Ε, σίγουρα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να βρούμε αυτές τις λύσεις, αυτά τα κίνητρα. Τελικά όμως πρόκειται για ένα πολιτικό έγγραφο που περιλαμβάνει πολιτικές δεσμεύσεις Δεν έχουμε όμως ε, κάτι το οποίο μπορούμε να επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη αν δεν ε, τηρούν τις δεσμεύσεις τους. Έτσι κι αλλιώς, τα πράγματα διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πραγματικά τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. να διευκολύνουμε αυτό που είπε η προηγουμένω όταν κάποιο ε, όντω ε, αποσπάται ε, και πηγαίνει σε μια αποστολή αυτό να λειτουργεί υπέρ του κατά την επιστροφή του και να μην θεωρείται χαμένο χρόνο. Έχουμε και αυτή τη διαδικασία ετήσια αναθεώρησης που θα πρέπει να εξετάσουμε όλα αυτά τα στοιχεία και να τα λάβουμε υπόψη, να δούμε τις βέλτες, τις πρακτικές να δούμε ποιος τα πηγαίνει καλύτερα. Αυτός είναι για μένα ο δρόμος από εδώ και πέρα. Συμφωνώ ότι είναι θέμα υλοποίηση στη τελική ανάλυση. Τώρα για την... Ε, Ευαισθησίας προς ε, συγκρούσεις, ε, Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την ανάλυση της σύγκρουσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το σύμφωνο όμως επισημαίνει ότι αυτό πρέπει να γίνεται όλο και περισσότερο και με τους συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να κάνουμε λοιπόν την ίδια ανάλυση των προβλημάτων της σύγκρουσης όταν σχεδιάζουμε την ε, απόκρισή μας. Για το ίδιο το σχέδιο δράσης λοιπόν, νομίζω ότι θα σταθούμε στην υλοποίηση του συμφώνου και της ενέργειες που απορρέουν από αυτό. Νέες διαδικασίε, πρόσληψης, κατάρτισης και το καθεξής. Δεν είναι ένα σχέδιο δράσης που προβλέπει ενέργειες επιτόπου, δηλαδή το πώς θα ανταποκριθούμε στη μετανάστευση. Θα, έχει, θα είναι ένα σχέδιο με προσδοτολισμό τη δράση. Σημειώνω βέβαια τα όσα είπατε, εντάσσονται σε μια ευρύτερη συζήτηση για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της μετανάστευσης. Όμως τελικά πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να συμβάλλουμε και εμέσως με χρηστή διακυβέρνηση, καλύτερες ε, δομές, ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου, σε όλες αυτές τις περιοχές από όπου προέρχονται οι μετανάστες, να συμβάλλουμε όσο μπορούμε για να μην φεύγουν από τις πατρίδες τους σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να βελτιώσουμε και την ε, διαχείριση των συνόρων, να δούμε την ε, ακτοφυλακή και το καθεξής. Σίγουρα πρέπει όμως να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συνεργασία. Το καινούριο στοιχείο εδώ είναι ότι πρόκειται για δέσμευση από τα κράτη-μέλη. Φυσικά δεν υπάρχουν κυρώσεις, υπάρχουν όμως μηχανισμοί υλοποίηση, ας πούμε. Αυτό δημιουργεί ένα πλαίσιο βελτίωση των πραγμάτων στο μέλλον. Για να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον ε, προπολογισμό και έπαμε με νέο πιο επικοινωνικό τρόπο. Με πολιετή σχεδιασμό και προβλέψεις και τελικά όλα αυτά έχουν να κάνουν και με το στρατηγικό προσανατολισμό. Κάποιες φορές θα πρέπει να έχουμε βραχυπρόθεσμες ε, ενέργειες. Συχνά όμως, αυτή η διαφορά που θέλουμε εμείς να πετύχουμε ε, γίνεται πιο μακροπρόθεσμα. είτε πρόκειται για το Σαχέλ, είτε για το κέρας Αφρικής, στη Μέση Ανατολή κτλ. Επομένω, προσπαθούμε να είμαστε ρεαλιστέ, να μην ε, βάζουμε ιδιαίτερα υψηλού, υπερβολικά υψηλού μάλλον στόχου. Έχουμε θέσει μα μια σειρά στόχων και ποσοτικών. Όμω, γενικά θέλουμε να επικεντρωθούμε, όπω και τα κατημέλη, στην ποιότητα, στι εθνικέ μεταρρυθμίσει και μετά από κοινού να έχουμε αποτελέσματα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βέβαια πρέπει να υπάρχει και ένα σύστημα μετά την ανάπτυξη δυνάμεων να μπορούμε να μετρήσουμε αυτό που κάναμε αν είχε κάποιον αντίκτυπο. Αυτά ευχαριστώ. Good luck. Uh, <laughs> Mr. Falek? Yes, just a quick reaction on two questions. Μία γρήγορη αντίδραση στις ερωτήσεις. Σε αυτό το οποίο είναι καινούριο. Ποια είναι τα όρια της μη στρατιωτικής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Το ίδιο ερώτημα θα ρωτούσα σε σχέση με την παγκόσμια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είχαμε όταν δεν την είχαμε. Η πρώτη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ήταν αποτελεσματική. Δεν ε, στάθηκε στο ύψος των προσδοκιών. Η δεύτερη στρατηγική τώρα δεν ξέρω αν θα σταθεί στο ύψος των προσδοκιών. Αν έπρεπε να επενδύσω ή να στοιχηματίσω σε αυτό, δεν θα έβαζα και πάρα πολλά χρήματα. Δεν θα πόνταρα στο ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει πιο ανθεκτικές τις κοινωνίες που βρίσκονται στην ευρύτερη γειτονιά μας, ούτε θα πόνταρα πολλά χρήματα στο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ένας πιο ασφαλής σε χώρο, σε 10 χρόνια από τώρα. Και σίγουρα δεν θα πόνταρα ότι θα αφαιρεθεί το μη στρατιωτικό σκέλος από αυτή την εξίσωση. Επομένως, βασική συνιστόσα της παγκόσμιας στρατηγικής που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό είναι ακριβώς αυτό. Και ο λόγος για τον οποίο έχουμε στρατηγικές και τις αλλάζουμε και εξελισσόμαστε και ε, από την πολιτική στήριξη πάμε σε νέα πολιτική στήριξη και σε νέο κείμενο. Είναι ο λόγος ότι δηλαδή είναι εξελικτικά, υψηλά εξελικτικό το διεθνές σύστημα και μερικές φορές είναι θέμα ταχύτητας. Δηλαδή νέες απειλές προκύπτουν ταχύτατα και ξαφνικά. Νέες προϋποθέσεις, νέες συνθήκες επικρατούν σε διάφορα πεδία μάχης, σε, διάφορα, ε, σε διάφορες αιστείες και όλα αυτά απειλούν την ασφάλεια της Υπήρου μας. Και γι' αυτό το στρατηγικό έγγραφο στόχο έχει να δώσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει αυτές τις νέες συνθήκες και νέες προϋποθέσεις. Όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Μολενάρ, ε, η μη στρατιωτική κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας έχει αποτελέσματα σε μακροπρόθεσμη βάση. Ο αντίκτυπος αυτού που κάνουν οι μη στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες φαίνεται σε μακροπρόθεσμη βάση και σε μερικές περιπτώσεις δεν φαίνεται και καθόλου. Δηλαδή δεν έχουμε τα αριθμητικά στοιχεία που ε, μας αποδεικνύουν τι θα συνέβαινε εάν δεν είχαμε αναπτύξει μία μη στρατιωτική κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα και αν δεν είχαμε, για παράδειγμα, δώσει δικαστική συνδρομή σε χ χώρα τη Αφρική ή ψη περιφέρεια. Δηλαδή, είναι εύκολο να δείχνει κανεί τα όρια τη μη στρατιωτική πολιτική ασφάλεια και άμυνα, και μάλιστα με το εφιστάμενο πλαίσιο. Είναι πολύ εύκολο εγχείρημα αυτό, πολύ εύκολη άσκηση είναι κανεί να δείξει τα όρια αυτή τη πολιτική. Όμω μην το υποτιμούμε, μην την υποτιμούμε. Μην την αφαιρέσουμε από τους στρατηγικούς υπολογισμούς που κάνουμε και από τη στρατηγική συζήτηση που λαμβάνει η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση την παγκόσμια στρατηγική μας. Ακριβώς διότι η δυνατότητα της ολοκληρωμένης, της ολοκληρωμένης προσέγγισης να υλοποιηθεί και να εφαρμοστεί 100% εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο η μη στρατιωτική συνιστόσα λειτουργεί και μπορεί να λειτουργήσει αντισταθμιστικά, να συμπληρώσει, να καλύψει κενά οι στρατιωτικοί στηρίζουν την ανάπτυξη μη στρατιωτικών μέσεων και άλλου είδους ε, αναπτυξιακές δράσεις επιτόπου και άλλου είδους συνδρομή όπως αυτή που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη διαχείριση των συνόρων και ε, για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Υπάρχουν δηλαδή περιορισμοί, τα μέσα ε, εξχεδιασμού τους έχουν κάποιους περιορισμούς και τα έγγραφα που συντάσσονται είναι περιοριστικά, δεν καλύπτουν τα πάντα, ωστόσο ε, θα ένιωθα πολύ λιγότερη εμπιστοσύνη εάν δεν τα είχαμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Άννα Πένφρατ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Να επανέλθω στο θέμα της απουσίας τελεχών. Στο career path, την επαγγελματική διαδρομή του υποψηφίου, υπάρχει αυτή η δυνατότητα αυτή είναι βεβαίως και ευθύνη των κρατών μελών. Τα αριθμητικά στοιχεία στο έγγραφο είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Δεν αποτελούσε αυτό μέρος των συζητήσεων πριν από λίγα χρόνια. Είναι δύσκολο να βρει κανείς αυτούς τους seconded officers. Και στις Βρυξέλλες πολύ συχνά μας λένε αν ας είμαστε φιλόδοξοι και θα βρούμε και στελέχη γιατί θα εμπλακούν τα κράτη-μέλη. Όμως, πολύ συχνά δεν εφαρμόζονται οι εντολές. Δηλαδή, στις Βρυξέλλες υπάρχουν σχέδια έκτακτης ανάγκης όταν δεν έχουμε την εμπειρογνωμοσύνη που είναι απαραίτητη για να υλοποιήσουμε την εντολή μας. Εάν δεν τα έχουμε αυτά, τι μπορούμε να κάνουμε την αποστολή που να είναι ρεαλιστικό και εφικτό. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες για τα νέα στοιχεία. Δεν είναι μόνο το περιβάλλον που αλλάζει, είναι και το γεγονός ότι αυτή η πολιτική είναι πολιτικό εργαλείο και εξαρτάται από τη δέσμευση των κρατών μελών, η πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Και γι' αυτό είναι χρήσιμο να βάζουμε τα κράτη-μέλη να σκέφτονται τι θέλουν να κάνουν με αυτό το εργαλείο θα πρέπει να δημιουργηθεί πολιτική όθηση, παρόλο που επί χάρτου οι διαφορές δεν είναι σημαντικές. Η διαδικασία είναι αυτή δηλαδή που θα κάνει τη διαφορά. Ένα τεχνικό ερώτημα να σας επευθύνω. Σε σχέση με το απαιτούμενο προσωπικό, ποια είναι η διαδικασία. Ένα άτομο, για παράδειγμα, που ταιριάζει στο προφίλ και στα χαρακτηριστικά, μπορεί να αυτοπροταθεί και μετά να πάρει άδεια από την υπηρεσία του και από το κράτος του. Ή πρέπει να περιμένουμε το κράτος μέλος να μας δώσει τον άνθρωπο να μας στείλει το συγκεκριμένο. Γιατί φανταζόμαι ότι υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι στα κρατημέλη που θέλουν είτε να κάνουν αυτή τη δουλειά, είτε να... Ε, ή και μόνο και μόνο για το επίδομα. Γιατί το ότι θα μετακινηθούν στο εξωτερικό έχει απολαβές και μπορεί να είναι αυτό αρκετό κίνητρο για αρκετούς, εκτός από τη φιλοδοξία. Και άλλοι έχουν απλά την φιλοδοξία Εν πάση περιπτώσει, χαριτολογώντας αυτά, ε, το ερώτημα παραμένει. Μπορεί να αυτοπροταθεί ο υποψήφιος ή πρέπει να περάσει από την ιεραρχία του πρώτα και το κράτος να τον προτείνει. Απάντηση. Κοιτάξτε, αυτό είναι δουλειά της CPCC. Τυπικά όμως νομίζω ότι τα κράτη-μέλη το κάνουν αυτό. Αν δεν υπάρχει όμως επαρκής υποψήφιος, έχουμε ορισμένε θέσει που είναι για προσωπικό που προσλαμβάνουμε. Και άρα εκεί μπορεί να μπει ένας εμπειρογνώμονα που να ταιριάζει με το προφίλ, με την περιγραφή, με το περίγραμμα εργασίας δηλαδή. Σταδιακά υπάρχει μεταστροφή από τους αποσπασμένους από τις κρατικές υπηρεσίες προς το προσωπικό που έχουμε προσλάβει επιτόπου με σύμβαση έργου. Υπάρχουν ειδικέ θέσεις στις αποστολές όπου θέλουμε να έχουμε εμπειρογνώμονες των κρατών μελών που να ε, είναι δημοσιοπάλληλοι. Έχουμε και τις δύο επιλογές, γιατί θέλουμε να αυξήσουμε τη συμμετοχή των κρατών μελών. Ο πρόεδρος, κοιτάξτε, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Εάν υπάρχει συμφωνία για μια συγκεκριμένη αποστολή, όλα τα κρατημέλη π.χ. έχουν συμφωνήσει για μια συγκεκριμένη αποστολή, Ακόμα όμως είναι φλού το ποιος θα τη φέρει σε πέρας. Δεν μπορούμε να έχουμε κάποιες διατάξεις σύμφωνα με τις πιες ε, τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να αρνηθούν ένα δικό τους δημόσιο υπάλληλο να μεταβεί άπαξ και αναγνωριστεί ότι ταιριάζει με το περίγραμμα εργασίας. Δηλαδή μπορεί το άτομο να αυτοπροταθεί και να πει «Κοιτάξτε τα προσόντα μου, μπορώ να είμαι υποψήφιος» και αν ναι, να μην αρνηθεί το κράτος μέλος, να τον αποσπάσει και να τον στείλει. Γιατί δεν θα έπρεπε το κράτος μέλος να παραπονεθεί κατά τη γνώμη μου, γιατί είχε συμφωνήσει να γίνει αποστολή. Από τη στιγμή που συμφωνεί να γίνει η αποστολή, κάποια στιγμή πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις του και όταν υπάρχει υποψήφιο και θεωρείται και κατάλληλο να μην τον αρνείται και να δέχεται να τον στείλει. Γιατί είναι θέμα ε, τήρησης υποχρεώσεων από πλευράς κράτους μέλους. Απάντηση. Μία από τις δράσεις είναι η αναθεώρηση, έτσι ώστε το κείμενο να είναι πιο ευέλικτο. Θα το αφήσουμε αυτό στους εμπειρογνώμονες. Καλώς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εάν δεν υπάρχουν ερωτήσεις από συναδέλφους, τότε να ευχαριστήσουμε τους τρεις εισηγητές για το ότι ήρθαν εδώ, για το ότι μας ενημέρωσαν για τις τελευταίες εξελίξεις σε μια πολύ επίκαιρη χρονική στιγμή σε σχέση και με τις χθεσινές αποφάσεις. Ας δούμε πώς θα γίνει η υλοποίηση και αν θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα σε αυτό τον κύκλο ζωής. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Λοιπόν. Ε, πάμε στο σημείο υπερτιμών 11 της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε την προσθέτηση μελέτη σε διαδικασία εφαρμογή σε Λευκή Βίβλος. Εμείς ζητήσαμε αυτή τη μελέτη μετά από την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε με τον Χαφιέ Σολάνα στις 16 Ιουνίου του 2016 και θελήσαμε να υπάρχει μια Λευκή Βίβλος για θέματα άμυνας. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να χαιρετήσω τον συγγραφέα το συντάκτη της μελέτης, Μέτρ Μωρό, ο οποίος ε, είναι ε, Εξοικειωμένο, ε, με την γαλλική λευκή βίβλο ε, και με γαλλικά προγράμματα. Ε, έχει εργαστεί για τις μόνιμες επιτροπές των ενόπλων δυνάμεων για θέματα στρατού στην Γερουσία της Γαλλίας. Έχει έναν μια πολύ καλή συνεργασία με εμπειρογνώμονες, με εκπροσώπους των κρατών μελών, με στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης και με το επιτελείο των το επιτελείο της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Έχουμε μπροστά μας τη μελέτη αυτή και με πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τις δικές σας τις προτάσεις και τα συμπεράσματά σας. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να παρουσιάσω τις βασικές μου ιδέες οι οποίες κινούνται γύρω από τρεις άξονες και ελπίζω να μην ξεπεράσω τα 20 λεπτά που μου έχουν δοθεί. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα χαρακτηριστικά των δύο διαδικασιών σχεδιασμού αμυντικής πολιτικής που υφίστανται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον, το NATO Defense Planning Process και την Ευρωπαϊκή Διαδικασία, η οποία δεν έχει συγκεκριμένη ονομασία και την οποία θέλω να αποκαλέσω με τον ίδιο τρόπο EUDPP, δηλαδή European Union Defense Planning Process. Αυτά καταρχάς, μετά θα σας παρουσιάσω τα θετικά και τα αρνητικά των δύο διεργασιών αυτών και στο τέλος θα προσπαθήσω να δώσω κάποιες πρόπτικες για την σύνταξη μιας λευκής βίβλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ευρωπαϊκή άμυνα. Ας ξεκινήσω με τα χαρακτηριστικά των δύο διαδικασιών και να μιλήσω πρώτα για το σχεδιασμό της άμυνας. Ο σχεδιασμός της άμυνας γίνεται με μια σειρά ερωτήσεων και λογικών απαντήσεων, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα εργαλείο αμυντικό, το οποίο ένα συγκεκριμένο έθνος ή μια συμμαχία θεωρεί απαραίτητο για να εκπληρώσει τις αμυντικές της φιλοδοξίες και να αντισταθεί στις ε, ε, επιθετικές απαντήσεις είναι μια διαδικασία η οποία εξαρτάται και από το κόστος και την προθεσμία κατασκευή στρατιωτικού εξοπλισμού. Να έχουμε εργαλεία αμυντικά που να αντιστοιχούν στις φιλοδοξίες και στις απειλές ε, που ε, έχει και που υφίσταται ένα συγκεκριμένο κράτος, έθνος ή μια συμμαχία. Εάν θέλετε να μιλάω πιο αργά, τότε θα μου δώσετε και λίγο παραπάνω χρόνο από τα 20 λεπτά. Ευχαριστώ. Επομένως, αναπόσπαστο στοιχείο για οποιαδήποτε διαδικασία αμυντικού σχεδιασμού είναι για τις πολιτικές αρχές η διατύπωση στόχων. Δηλαδή, περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται περί διαχείρισης κρίσεων στη γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για την εγγύηση της ασφάλειας της ευρωπαϊκής επικράτειας. Δεν θα φτιάξουμε τα ίδια αμυντικά εργαλεία και για τη μία και για την άλλη περίπτωση, αλλά διαφορετικά. Σημαντικό είναι να έχουμε υπόψη μας το εξή. Όπως και αν ονομάσουμε αυτό το στοιχείο το κατεξοχήν πολιτικό, είτε το πούμε λευκή βίβλο, είτε το πούμε αμυντική στρατηγική ή στρατηγικές έννοιες και ιδέες. Ο αμυντικός σχεδιασμός αυτό καθεαυτός δεν μπορεί να ξεκινήσει χωρί αυτή τη λευκή βίβλο, και αν γιατί, Γιατί αν δεν ξέρετε τι θέλετε να χτίσετε, ε, δεν θα καταφέρετε να το χτίσετε. Είναι σαν να χτίζετε σπίτι. Δεν μπορείτε να φτιάξετε σπίτι χωρίς σχέδιο. Είναι πολύ πιο δύσκολο αυτό. Επομένως, θα ήθελα να σας περιγράψω τις δύο αυτές διαδικασίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ε, κατά αντιπαραβολή, ε, υπογραμμίζοντας τις ομοιότητες και τις διαφορές. Αριστερά, λοιπόν, έχουμε το, του ΝΑΤΟ και δεξιά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από πότε υπάρχουν. Η διαδικασία η νατοϊκή ε, στρατηγικού σχεδιασμού είναι ήδη 50 ετών. Είχαμε το Defense Planning Review του 71 κείμενο. Είναι μια διαδικασία πολύ καλά εδρωμένη, τα κράτη την έχουν συνηθίσει και την ξέρουν και παρόλο που θεωρείται επαχθής και γραφειοκρατική, γίνεται αποδεκτή από τα κράτη χάρη στη δύναμη της συνήθειας. Έχει υποστεί βασικό ανασχεδιασμό και αναδιαμόρφωση το 2009 και έχει γίνει πολύ πιο αποτελεσματική από ό,τι στο παρελθόν. Όμως η ευρωπαϊκή διαδικασία στη δεξιά στήλη είναι πολύ πιο πρόσφατη, είναι 15 ετών και όχι 50, υλοποιήθηκε και καταρτίστηκε σε τρία στάδια. Από το 1999 μέχρι το 2005 ήταν το πρώτο στάδιο, το στρατιωτικό σκέλος υπό την ευθύνη της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης CMEU με τη βοήθεια του ε, Γενικού Επιτελείου ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τελικά δημιουργήθηκε ένας μηχανισμός ανάπτυξης ικανοτήτων CDM, Capacity Building Mechanism. Μετά έχουμε τη δεύτερη φάση της άμυνας. Υπό την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια από το 2005 και μετά και έχουμε το CDP, τρίτο στάδιο είναι το στάδιο που ξεκίνησε το 2016 και έχει να κάνει με ε, το ετήσιο έλεγχο των αμυντικών θεμάτων, QUAD, και τις διάφορες πρωτοβουλίες. Πέσκο, έργων Πέσκο. Θα ήθελα τώρα να σας παρουσιάσω το γενικό προσανατολισμό κάθε μίας από αυτές τις δύο διαδικασίες. Η νατοική διαδικασία ε, δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου για να έχουν οι σύμμαχοι τις απαραίτητες δυνατότητες να υπερασπιστούν τη συμμαχία. Αυτός ήταν ο βασικός σκοπός και γι' αυτό και καλύπτει το σύνολο του φάσματος των στρατιωτικών εξοπλισμών. Αντιθέτως, η ευρωπαϊκή διαδικασία έχει να κάνει με την κοινή εξωτερική πολιτική που και πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Στόχος του ΠΕΣΚΟ και των λοιπόν εργαλείων είναι να δώσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ικανότητα αυτόνομης δράσης για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαχειριστεί τις κρίσεις στην ευρύτερη της γειτονία. Το 2000 ε, ε, όμως 18 απομακρυνθήκαμε γιατί η τελευταία εκδοχή του κειμένου καλύπτει το σύνολο του φάσματος του στρατιωτικού εξοπλισμού και γίνεται λόγος για τη στρατιωτική κινητικότητα, κάτι το οποίο απέχει από, την αρχική, από τον αρχικό σχεδιασμό. Τρίτο σημείο σύγκριση είναι το επιχειρησιακό σκέλο. Η νατοική διαδικασία είναι προσανατολισμένη προ τα αποτελέσματα και αυτό είναι απολύτω κατανοητό γιατί κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου έπρεπε η συμμαχία να έχει τι δυνατότητε και τα μέσα τα οποία θεωρεί ότι χρειάζεται. Και γι' αυτό έχουμε τρία βασικά χαρακτηριστικά στον, στην, στην νατοική διαδικασία. Top-down, από πάνω προ τα κάτω. Είναι πολύ καθ κατευθυντική και διευθυντική. Δίνει ένα κατάλογο με ψώνια που πρέπει να κάνει το κράτος μέλος. Ε, το κάθε κράτος ε, μέλος ενίοτε και χωρίς να το θέλει βάσει του κανένα consensus minus one, συνένεση μείον ένας. Είναι μια διαδικασία κυκλική που κρατάει τέσσερα χρόνια και επαναξιολογούμε το αμυντικό σχέδιο σε σχέση με τις απειλές κάθε τέσσερα χρόνια. Είναι μια διαδικασία αρκετά ε, διεισδυτική γιατί πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν τις δυνατότητες που τους ζητούμε να έχουν και ότι έχουν κάνει τα ψώνια που τους χρειάζεται και που τους ζητούμε να κάνουν. Όμως η ευρωπαϊκή διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαφορετική. Θέλουμε να βρούμε τομεί πάνω στους οποίους τα κράτη-μέλη είναι έτοιμα να συνεργαστούν. Έχουμε τρία χαρακτηριστικά αντίστροφα από την ατοική. Έχουμε top-down στο στρατιωτικό σκέλος και bottom-up από κάτω προς τα πάνω από την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Αμυντική Υπηρεσία. Ο καθένα εκπληρώνει τι ε, υποσχέσει του εάν το επιθυμεί και το αποτέλεσμα αξιολογείται συλλογικά δεν έχουμε naming and shaming, δεν έχουμε ατομική επίρρηψη ευθυνών στο χ υψη κράτος. Η διαδικασία δεν είναι κυκλική, ε, ξεκινάει μόνο αν το ανακηρύξει το Συμβούλιο και το θεωρήσει αυτό χρήσιμο και δεν είναι διεισδυτική, ε, δηλαδή καλεί τα κρατημέλη να παίξουν το παιχνίδι, δεν τα ελέγχει κατά πόσο το έπαιξαν και γιατί δεν το έπαιξαν καλά. Τώρα, από πλευράς ΝΑΤΟΥ είναι μία και μόνη οργάνωση, η οποία έχει και την ευθύνη. Το ΝΑΤΟ. Βεβαίως, εκεί επισέρχονται πολλές διαφορετικές και υπηρεσίες. Έχουμε τα δύο στρατιωτικά επιτελεία, τη Στρατιωτική Επιτροπή και τη Διεθνή Γενική Γραμματεία, με ένα τμήμα το οποίο έχει αναλάβει την διαδικασία, σημειώνει τις επενδύσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα και ε, είναι σημαντικές. 350 άτομα στο σύνολο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε έξι φορείς που επισέρχονται εκεί. Για το CDP έχουμε την EUT, άλλον οργανισμό για το CPM, άλλη υπηρεσία για την ΠΕΣΚΟ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει τη γραμματεία του ΦΕΔ, και έχουμε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που προσδιορίζει το ύψο των φιλοδοξιών μα. Πολλοί και διαφορετικοί φορεί λοιπόν, αλλά πολύ λίγο το προσωπικό. Περίπου 30 άνθρωποι ε, εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία και στου έξι αυτούς φορείς ή στα αυτού φορεί Η νατοική πώ λειτουργουν αυτέ οι δυο διαδικασίε, η νατοικη διαδικασια περιγραφεται σε όλε τι λεπτομέρειε ένα έγγραφο όχι υψηλή ταξινόμηση, το οποίο κυκλοφορεί εντό τη συμμαχία. Εκεί υπάρχουν και τα βασικά ε, για τη διαδικασία τα οποία μπορεί κανείς να βρει και στο διαδίκτυο ελεύθερα. Ε, τα κράτη-μέλη εμπλέκονται ιδιαίτερα σε αυτή τη διαδικασία. Όμως η ευρωπαϊκή διαδικασία είναι πολύ πιο δύσκολο να την προσεγγίσει κανείς γιατί αποτελεί το άθροισμα των διαφορετικών ικανοτήτων και διαδικασιών απόκτησης ικανοτήτων που έχει το κάθε κράτος μέλος τα κράτη-μέλη προσδίδουν πολύ λιγότερη σημασία στην ευρωπαϊκή διαδικασία από ότι στην ατοική. Έχουμε μικρά κράτη-μέλη που δεν έχουν τους απαραίτητους ανθρωπίνους πόρους για να παρακολουθήσουν και τις δύο διαδικασίες ταυτοχρόνως και γι' αυτό παρατούν την ευρωπαϊκή και επιλέγουν την ατοική διαδικασία. Να σας δείξω πώς λειτουργεί σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια. Για την ατοική διαδικασία κάθε κύκλος αποτελείται από πέντε ε, φάσεις. Πρώτη φάση είναι πολιτική προσταγή. Είναι το πράσινο κομμάτι που βλέπετε στο κέντρο του κύκλου. Αυτές οι πολιτικές διρεκτίβες και οδηγίες μεταφράζουν σε στρατηγικούς όρους τους στόχους της συμμαχίας όπως αναγράφονται στις συνθήκες και αυτά τα εξετάζει το στρατηγικό κόνσεπτ που το τελευταίο είναι το 2010 και επικυρώνονται στις συνόδους κορυφής του ΝΑΤΟ. Είχαμε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ μία φορά κάθε δύο χρόνια. Στη συνέχεια έχουμε τη φάση όπου καταρτίζεται ο ελάχιστος κατάλογος απαραίτητων ικανοτήτων για να ικανοποιηθεί η φιλοδοξία ε, η στρατιωτική και η πολιτική. Τρίτη φάση είναι να δοθούν στόχοι για κάθε μέλος της συμμαχίας. Τέταρτη φάση, υλοποίηση των αποφάσεων ανάθεση στόχων είναι το, ο δακτύλιος ο μπλε που βλέπετε. Και πέμπτη και τελευταία φάση είναι η εξή. Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, ε, αναθεώρηση του δυναμικού των ικανοτήτων που γίνεται κάθε δύο χρόνια και που έτσι γίνεται παρήθμιση και κατάλογος απογραφή των διαθέσιμων δυνάμεων. Μιλούμε για όλες τις σημαντικές δυνάμεις, όχι αυτές που μπορούν να αναπτυχθούν σε επίπεδο ΝΑΤΟ, αλλά και τις λοιπές δυνάμεις μιας χώρας. Τώρα, στην ευρωπαϊκή διαδικασία τα πράγματα είναι κάπως πιο περίπλοκα. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε τη λογική που ακολουθεί ε, μια πυραμίδα, ένα σιλό, μια μεγάλη δεξαμενή. Πρώτη στήλη, το CDM έχει συγχωνευτεί με το CDP. Στη δεύτερη στήλη έχουμε το ΠΕΣΚΟ που είναι ε, κρατική εθνική αρμοδιότητα και στην τρίτη στήλη έχουμε αυτά που, για τα οποία έχει αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλοι λοιπόν καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι ο συντονισμός για όλα αυτά τα διακυβεύματα και πόσο το πρόγραμμα εργασιών της ΦΕΔ, εκεί που υπάρχουν τα χρήματα δηλαδή, μπορεί να συνδεθεί με ένα σοβαρό αμυντικό σχεδιασμό. Εάν τώρα δούμε πώς ε, διαρθρώνεται το CDM με το CPM, εδώ αυτό είναι το αποτέλεσμα της διάρθρωσης της αριστερής στήλη, της αριστερής αν θέλετε δεξαμενής της προηγούμενης διαφάνειας. Μπορώ να επεκταθώ αν θέλετε για το θέμα αυτό. Τώρα για τις αδυναμίες των δύο αυτών διαδικασιών. Καμία από αυτές τις διαδικασίες δεν επέτρεψε να εκπληρωθούν οι φιλοδοξίες ούτε του ΝΑΤΟ ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Μωρίς Λαγκλουά και άλλοι Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες το 2014 εκτιμούσε ότι η, Νατοϊκή Συμμαχία εκπληρώνει μόνο το 14% των φιλοδοξιών της και κατά 5% χάρη στη συνεισφορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατά προσήγηση ε, το ίδιο ε, πρέπει να είναι το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εκπληρώσει τις φιλοδοξίες της για τις πιο απαιτητικέ αποστολές έτσι όπως χαρακτηρίζονται από τις συνθήκες, δηλαδή για την επιβολή της ειρήνης, την ειρηνευτική διαδικασία. Ωστόσο, ε, οι διαδικασίες αυτές έχουν άλλες αρετές, εξού και είναι απαραίτητες. Είναι η σπονδυλική στήλη της Νατοικής Συμμαχίας ο αμυντικός σχεδιασμός και η διαδικασία αυτή. Και γι' αυτό το λόγο περιγράφεται ως το, ως το συνδετικό ιστό την κόλλα που ενώνει τα μέλη της συμμαχίας μεταξύ τους. Περιγράφεται ως το καλούπι για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ ευρωπαϊκών και αμερικανικών στρατιωτικών και άλλων δυνάμεων. Ποιος κάνει τι. Είναι ένα στρατηγικό ερώτημα εντός της νατοικής συμμαχίας. Το... Στο EUDPP στο στρατηγικό σχεδιασμό των αμυντικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα ότι υπάρχει βούληση για ανεξάρτητη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια πλατφόρμα για να συνεργαστούν περισσότερο τα κράτη-μέλη μεταξύ τους εάν το επιθυμούν άρα είναι σωστό συνομιλητής της βιομηχανίας του κλάδου και απαντά σωστά στα ερωτήματα πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα η νατοική διαδικασία μεταλαμπαδεύει την αμερικανική νοτροπία, δεν επιδέχεται πολλές ε, κριτικές, ε, εξαρτάται από όλες τις αμερικανικές στρατηγικές και έχουμε ε, και κατά κύριο λόγο κατεξοχήν τους αντιβαλιστικούς πυράβλους, τους αμυντικούς, δηλαδή βασικό αμερικανικό δόγμα και γι' αυτό κατηγορείται καλός ή κακός ότι ενθαρρύνει την αμερικανική στρατιωτική βιομηχανία. Η ευρωπαϊκή τώρα διαδικασία δυστυχώς ε, οδήγησε στην ανάπτυξη λίγων ικανοτήτων, μικρών ή και καθόλου τα τελευταία 15 χρόνια. Έχει σημαντικά σφάλματα η ευρωπαϊκή διαδικασία. Δεν είναι ειλικρινείς οι δηλώσεις πολλών κρατών μελών. Δεν εμπλέκονται ε, ενεργά, δραστήρια και διαπράττουν η ευρωπαικη διαδικασια δεν ειναι ειλικρινη οι δηλώσει λογικής και έτσι είναι μη επιχειρησιακά αυτά που κάνουν και μη λειτουργικά. Η ΦΕΔ και η ΠΕΣΚΟ είναι εργαλεία πολύ πρόσφατα και δεν μπορούμε να τα κρίνουμε. Σε δέκα χρόνια θα μπορέσουμε να έχουμε τη διάβγεια και την απαραίτητη αντικειμενικότητα για να κρίνουμε την αποτελεσματικότητά τους. Έρχομαι τώρα στις πιθανές εξελίξεις και κάποια σημεία προβληματισμού για το μέλλον. Θα απέκλεια το ενδεχόμενο της μοναδικής διαδικασίας ε, δεν πρόκειται να εξαφανιστεί ο αμυντικός σχεδιασμός του ΝΑΤΟ παρά μόνο να εξαφανιστεί και η ΝΑΤΟϊκή συμμαχία. Και αυτό το ενδεχόμενο φυσικά αποκλείεται γιατί η διαδικασία αμυντικού σχεδιασμού είναι και η σπονδυλική στήλη του ΝΑΤΟ. Αποκλείεται λοιπόν να εξαφανιστεί ό,τι και αν λέει και ό,τι και αν κάνει ο πρόεδρος Τραμπ. Ωστόσο η ευρωπαϊκή στρατηγική ε, πρέπει να έχει φιλοδοξία και το ελάττωμά της είναι ότι δεν έχει αρκετή φιλοδοξία. Για να γίνει θα πρέπει να τροποποιηθούν οι συνθήκες ή να μην εφαρμοστούν. Άρα, μπορεί κανείς να διανοηθεί τη συγχώνευση αυτών των δύο διαδικασιών. Η απάντηση είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε ίδιο αμυντικό εργαλείο με, ε, όταν έχουμε αμερικανικές δυνάμεις, τουρκικές, καναδέζικες, βρετανικές και άλλες. Δηλαδή όταν έχουμε τόσο ετερόκλητες χώρες δεν μπορούμε να έχουμε ένα και μόνο ενιαίο αμυντικό εργαλείο ίδιο για όλους. Άρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βραχυπρόθεσμα, μπορούμε να υιοθετήσουμε διάφορα μέτρα. Καταρχάς, να περιγράψουμε πολιτική οδηγία που θα εκφράζει στο στρατιωτικά τους αμυντικούς στόχους που επιθυμεί το Συμβούλιο. Συντάχθηκε το κείμενο στα τέλη του 2016 και δεν λαμβάνει υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και γιατί το κάνει αυτό, διότι τα κράτη-μέλη θέλησαν να εκφράσουν ένα φιλόδοξο στόχο, δηλαδή το στόχο της προστασίας της Ένωσης και των πολιτών της, όχι μόνο εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας δηλαδή, αλλά δεν εξέτασαν τι αυτό συνεπάγεται στην πράξη. Το ανέθεσαν αυτό στους στρατιωτικούς να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. Οι στρατιωτικοί έκαναν ό,τι μπορούσαν, αλλά δεν μπορούσαν να υποκαταστήσουν πλήρως τους πολιτικείς. Άρα, κατέληξαν στην κατασκευή ενός εργαλείου για αυτή την ε, ευρωπαϊκή ε, πολιτική, όχι στο να προστατεύσουν την Ένωση από τους δικούς της τους ίδιους πολίτες. Πρόκειται για κενά των κρατών μελών, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κενά που έπρεπε να καλυφθούν ε, θα χρειάζονταν όχι τα 13 δις που έβαλαν πάνω στο τραπέζι, αλλά περίπου 100 δις για να καλυφθούν τα κενά των κρατών μελών. Αν θέλουν δηλαδή να ανταποκρίνονται οι πράξεις ε, με τα λόγια τους, τα κράτη-μέλη θα πρέπει ή να δώσουν μέσα που να αντιστοιχούν στο ύψος των φιλοδοξιών τους ή να μειώσουν τις φιλοδοξίες τους στο ύψος των μέσων που διαθέτουν. Είναι αυτοί οι δύο τρόποι, οι μόνοι τρόποι να συγγράψει κανείς μια λευκή βίβλο. Αν έχουμε τεράστιες φιλοδοξίες και πολύ λίγα μέσα, τότε ε, το πληρώνουμε γιατί χάνουμε την αξιοπιστία μας. Δεν μπορεί αυτά τα δύο δηλαδή να αποκλίνουν. Πρέπει να κινούνται στο ίδιο επίπεδο, υψηλό ή χαμηλό, όποιο και αν είναι αυτό. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να πω και το εξής. Στη διαφάνεια βλέπουμε το, το κόκκινο τετράγωνο στο κάτω μέρος της οθόνης, το Φεβρουάριο του 2019 θα συγγραφούν οι νέες πολιτικές οδηγίες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Θα είναι πολύ δύσκολο να περιγραφεί ένα νέο επίπεδο στρατιωτικών φιλοδοξιών σε έτος ευρωεκλογών. Άρα να ξεκινήσουμε από το υφιστάμενο επίπεδο και να συγχρονίσουμε ό,τι μπορούμε να συγχρονίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 19 που είναι έτος εκλογών. Δηλαδή να γίνει κυκλική η ευρωπαϊκή διαδικασία και να συγχρονιστεί με την ατοική διαδικασία ε, οι αντίστοιχοι φορείς και υπηρεσίες εργάζονται εδώ και ε, αρκετό καιρό και δεν θα ήταν ευγενικό να ε, προστρέξω εγώ να τους πάρω τη θέση και να σας αποκαλύψω δουλειά που κάνουν ήδη εκείνοι. Επιπλέον, δεν είναι λογικό να ζητούμε από τους 30 ανθρώπους που ασχολούνται αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο να κάνουν την ίδια δουλειά με τους 350 ανθρώπους που κάνουν την αντίστοιχη δουλειά στο πλαίσιο της Νατοικής Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Δεν είναι αυτό δίκαιο και είναι πολύ δύσκολο όλη αυτή η διαδικασία να συγγραφεί σε ενιαίο έγγραφο, το οποίο όμως ποιον θα έχει συγγραφέα. Κάθε υπηρεσία και φορέα θα θέλει να έχει αυτή τα πρωτεία και να λέει ότι αυτή το συνέγραψε. Ε, υπάρχει δηλαδή και αυτή η δυσκολία και αυτό το ακαθόδε σημείο. Για τη λευκή βίβλο το βασικό για μένα δεν είναι το κατά πώς θα πρέπει να γραφτεί μια λευκή βίβλος ή όχι. Είναι απαραίτητο γρανάζει δεν μπορεί να υπάρξει διαδικασία σχεδιασμού χωρίς λευκή βίβλο. Το θέμα είναι πότε πρέπει να γραφτεί και πώς. Για το πότε λοιπόν θα πρέπει να εγκριθεί σε, με ορίζοντα το 2021 για να γίνει ταυτόχρονα ο κύκλος ο ευρωπαϊκός με τον κύκλο τον ατοϊκό ο οποίος θα ξεκινήσει το 2023. Άρα μετά τις εκλογές του 19 ή και πριν περιμένουμε τις εκλογές θα μπορούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συζητήσει έναν οδικό χάρτη πιο, πιο συγκεκριμένο και στις ακροάσεις των μελλοντικών επιτρόπων και του μελλοντικού είπα του εκπροσώπου για θέματα εξωτερικής πολιτικής να τεθούν όλα αυτά τα θέματα για να μην χάσουμε χρόνο. Ε, ε, δεν είναι ανέφικτο αυτό το εγχείρημα. Σίγουρα δεν θα είναι μια λευκή βίβλος αλλά γαλλικά ή αλλά αγγλικά. Δεν θα είναι ένα έγγραφο 100 σελίδων με πάρα πολλές λεπτομέρειες που να περιλαμβάνει τους αμυντικούς στόχους ε, σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε στρατιωτικό. Δεν μπορεί να είναι κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε όμως να είναι μια λευκή βίβλος η οποία να απηχεί το στρατηγικό κόνσεπτ όπως κάνει και το ΝΑΤΟ, περίπου 10 σελίδες δηλαδή και να περιγράφει τους αμυντικούς στόχους. Είναι κάτι το εφικτό που μπορούν να το κάνουν τα κρατημέλη. Το έκαναν και το 2016 όταν υιοθέτησαν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για ε, το σχέδιο υλοποίηση τη Παγκόσμια στρατηγική Και το κάνουν κάθε φορά που θετούν μια πολιτική οδηγία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, τη Βορειοατλαντική Συμμαχία, Να εμπνευστούμε δηλαδή από αυτό που γίνεται ε, στο ΝΑΤΟ. Οι πολιτικοί στόχοι να αποστασιοποιηθούν από τους στρατιωτικούς στόχους και άπαξ και οθετηθούν οι πολιτικοί στόχοι να ζητηθεί από τη Στρατιωτική Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις που να συνάδουν με τους πολιτικούς στόχους και στη συνέχεια να τροποποιηθούν οι προτάσεις αυτές σε πολιτικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ κοντά στη συγγραφή ε, ε, μιας λευκής βίβλους. Είναι κρίμα που το 2016 δεν μπορέσαμε να φτάσουμε ε, στο τέλος και πλησιάσαμε τόσο κοντά. Εφόσον δεν υπάρχει λοιπόν το κοινό πλαίσιο σε σχέση με τον ΝΑΤΟ, πρέπει ωστόσο να ε, προχωρήσουμε προς ένα ενιαίο οδικό χάρτη και όχι να έχουμε 5-6 διαφορετικούς όπως έχουμε τώρα. Τέλος, θεωρώ ότι επιβάλλεται μία μεταρρύθμιση της πολιτικής είτε ε, για να έχουμε μία νέα προσέγγιση ε, που θα εξοικονομήσει πόρους για την Ένωση. Ε, θα έχουμε έτσι μια πιο ενιαία προσέγγιση στην ε, αμυντική πολιτική, είτε να έχουμε ένα πραγματικό ερευνητικό οργανισμό σαν έναν ευρωπαϊκό DARPA. Κλείνοντας, μπορώ να πω ότι η διαδικασία σχεδιασμού της αμυντικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αναποτελεσματική και πολύ περίπλοκη αυτή τη στιγμή. Δεν δημιουργεί κάποια ικανότητα από το που δημιουργήθηκε και υπάρχει σημαντικός κίνδυνος παρόλες τις προσπάθειες και πρωτοβουλίες που έχουν ξεκινήσει το 2016 να παραμείνουν επί χάρτου. Μέχρι τώρα τα κράτη-μέλη ε, έχουν ακολουθήσει αυτή την άγουσα γιατί πολύ απλά δεν θέλουν να έχουν επιπρόσθετο κατάλογο ε, προϋποθέσεων και όρων που θα πρέπει να πληρούν. Με το κοινό ταμείο Άμυνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση όμω θα ε, δώσει σημαντική χρηματοδότηση. Πρέπει να δώσουμε βέβαια πόρους ε, στον κλάδο, αλλά με κριτήρια. Ε, και για να γίνει αυτό πρέπει να βελτιώσουμε το σχεδιασμό. Αν οι Ευρωπαίοι ηγέτε θέλουν πραγματικά μια Ευρώπη που προστατεύει, αν εσείς ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανταποκριθείτε θετικά ε, σε αυτό το ερώτημα, πρέπει να απαντήσετε και στο εξή ερώτημα. Με τι ακριβώς θα γίνει αυτό, με ποια μέσα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σα και είμαι στη διάθεσή για τυχόν ερωτήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας είπατε, για την επισκόπηση, την ανάλυση, τις ε, προτάσεις. Νομίζω ότι κανονικά ε, θα έπρεπε πρώτα να τα αφήσουμε έτσι λιγάκι να κάτσουν, όπως λέμε χαρακτηριστικά. Να κάτσουν λοιπόν όλες αυτές οι πληροφορίες, ε, να τα διαβάσουμε μόνοι μας. Και μετά ε, θα μπορούσαμε να έχουμε την ευκαιρία να υποβάλουμε τις ερωτήσεις μας. Αλλά έχω την εντύπωση ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε καλύτερα εάν ε, λάβουμε ε, κατά λέξη τα κράτη-μέλη και ζητήσουμε αυτό το οποίο κατ' ουσίαν έχουν ήδη δηλώσει σε επίπεδο αρχής. Δηλαδή διαδικασίες όπως είναι η διαδικασία CAD, αυτές οι διαδικασίες να τις λάβουμε ως ένα μοχλό και να πούμε, ξέρετε κάτι, ξέρετε τώρα τι έχουμε, εξ αυτών μπορούμε να ορίσουμε το τι χρειαζόμαστε και παρακαλώ ε, λειτουργήστε, αντιδράστε, συγκεντρώστε τους εμπειρογνώμονές σας και πάρτε και τα χρήματα που σας διαθέτουμε έτσι ώστε σε τέτοιου είδους διαδικασίες να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι τέτοιου είδους ε, μελέτες ε, θα πρέπει να τις διαθέσουμε και στους ε, συναδέλφους μας στα Εθνικά Κοινοβούλια για να μπορέσουν και αυτοί να μελετήσουν αυτές τις μελέτες και να τις συμπεριλάβουν στις τοποθετήσεις τους και επίση και για να μπορεί κάθε προεδρία να έρχεται αντιμέτωπη με αυτές τις ε, μελέτες για να γνωρίζει και αυτή το τι ισχύει και τι είχε αποφασιστεί εδώ και χρόνια. Και επίση το τι δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα. Βλέπω ότι ο συνάδελφος Τρογεύσκη ζητάει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την παρέμβαση. Σπανίως έχουμε τόσο επικριτικές ε, παρουσιάσεις. Έχω ορισμένες παρατηρήσεις ε, και ένα ερώτημα. Πράγματι, έχουμε πολλά έγγραφα και οι πραγματικές ε, και απτές αποφάσεις λείπουν. και σε ό,τι έχει να κάνει με την ε, άμυνα και την ασφάλεια είναι μια σημαντική επίκριση, αλλά αληθής. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια στο Κοινοβούλιο έχω δει πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα εδώ. Δεν βλέπαμε το ζήτημα της ε, ασφάλειας παλιά. Ενώ τώρα αναγνωρίζουμε ότι είναι σημαντική η ασφάλεια. Επιπλέον, οι πόροι προηγούνται τη απόφαση. Τώρα έχουμε την απόφαση τη Επιτροπή και του Συμβουλίου για την αύξηση της χρηματοδότησης για τον τομέα τη ασφάλεια. η καταπολέμηση των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, ε, η χρηματοδότηση κοινών ενεργειών, χρηματοδότηση του στρατού μέσω της έρευνας. Έχω λοιπόν δύο ερωτήσεις. Βλέπουμε πράγματι αλλαγές σε ό,τι αφορά την προσέγγιση ως προς την ε, λήψη πολιτικών αποφάσεων. Έχει αλλάξει κάτι λοιπόν στην ατμόσφαιρα για την ε, λήψη πραγματικών αποφάσεων. Και δεύτερον, αυτή η έλλειψη βούλησης για την ε, ανάληψη συγκεκριμένης δράσης, τι μορφή παίρνει, πού βλέπουμε δηλαδή πραγματικά αυτή την έλλειψη ε, βούλησης, αυτή την αδράνεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άλλες ερωτήσεις παρακαλώ. Από ό,τι βλέπω ε, δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Ως εκ τούτου σας δίνω το λόγο για να απαντήσετε. Πράγματι, από το 2016 υπήρξε μια σημαντική αλλαγή στο ευρύτερο κλίμα ε, με βάση διάφορους παράγοντες που τους γνωρίζετε όλους, δεν χρειάζεται να τους επαναλάβω εδώ. Γενικά η νοοτροπία, το mindset που λέμε στα αγγλικά, έχει αλλάξει δραματικά. Και αποδεσμεύτηκε μια σημαντική ποσότητα ενέργειας στον τομέα της ε, άμυνας που οδήγησε σε μια σειρά ενέργειες Επομένω, ε, υπάρχει μια σημαντική έτσι, αλλαγή, ε, μια νέα ενέργεια. Πρέπει όμω αυτή να τη διατηρήσουμε και να την εστιάσουμε για να γίνει αποτελεσματική. Ιδάλω θα έχουμε ε, διάφορες πρωτοβουλίες που δεν θα έχουν μια στόχευση που θα φέρει τα απαραίτητα αποτελέσματα. Όλες οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να τις συνδέσουμε καλύτερα, να τις κάνουμε πιο αποτελεσματικές. Πρέπει λοιπόν να διαμορφώσουμε τι απαραίτητε διασυνδέσει μεταξύ ευρωπαϊκού, εθνικού επίπεδου. Ιδάλλως, όλες αυτές οι πρωτοβουλίε θα μείνουν επί χάρτου, όπως είχε γίνει παλιότερα. Και αυτό θα είναι καταστροφικό, γιατί θα ε, δώσουμε την εντύπωση, θα δώσετε μάλλον την εντύπωση στου Ευρωπαίου πολίτε ότι ε, ε, ασχολείστε με αυτό το ζήτημα, ότι ε, θέλετε την Ευρώπη που προστατεύει, αλλά στην πράξη θα δούμε ότι αυτό δεν ισχύει. Η Ευρώπη δεν λειτουργεί, θα σα πούν. Γι' αυτό πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Δεν μπορούμε, κύριε Πρόεδρε, παρότι και με κάθε σεβασμό, δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πράγματα ε, να προχωρήσουν έτσι. Πρέπει, ε, αντιθέτως, να υπάρχει αυξημένη επαγρύπνηση. Και αυτό, με αυτό περνώ στο δεύτερο ερώτημα. Η έλλειψη βούλησης που εντοπίζεται μέσω, για παράδειγμα, του, σχεδιασμού, του αμυντικού σχεδιασμού. Αν δεν υπάρχει αμυντικό σχεδιασμό, αν δεν είστε σε θέση εσεί, οι Ευρωπαίοι ηγέτε, εσεί, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ε, διατυπώσετε του αμυντικού σα στόχου, να κάνετε αυτή την περίφημη λευκή βίβλο, που λέτε ότι θέλετε τόσο πολύ από το 2016. Ε, στην έκθεση μπορείτε να βρείτε σε παράρτημα όλες οι εκθέσεις και τα ψηφίσματα που έχετε εκδώσει από το 2016 αν κάνετε απλώ δεήσει, αυτό δεν πρόκειται να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Πρέπει να περάσετε στην πράξη και στη δράση. Στι επόμενε ευρωεκλογέ, λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένε δεσμεύσει, ε, με τι οποίε θα επιφορτήσετε και τον επόμενο επίτροπο, για παράδειγμα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτε μέχρι τώρα γιατί δεν έχουν δώσει μια λευκή βίβλο, γιατί έχουν κατά νου μια ε, λευκή βίβλο όπως κάνουμε στη Γαλλία, που ξεκινάει με, ένα, με μια παρήθμιση των ε, κινδύνων και καθώς δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε μια παρήθμιση αυτών των κινδύνων χωρίς να σφαχτούμε, λέμε «Α, είναι πολύ επικίνδυνο, μην το κάνουμε καθόλου». Όμω μπορούμε να κάνουμε μια διαφορετική λευκή βίβλο. Όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λέει «Θέλω να είμαι σε θέση να διαχειρίζομαι εξωτερικούς κινδύνους», να ενισχύω τους εταίρους και να προστατεύω την Ευρωπαϊκή Άμυνα, ε, Ένωση Άμυνας είναι κάτι το εξαιρετικό. Για πρώτη φορά θεσπίζει και θέτει αμυντικούς στόχους. Τώρα πρέπει όλα αυτά βέβαια να μπορέσουμε να τα μεταφράσουμε σε κάτι πιο συγκεκριμένο που να μπορούν να κατανοήσουν οι στρατιωτικοί και να μπορούν να αρχίσουν τον ε, πρακτικό σχεδιασμό. Διαφορετικά θα γίνει μια διασπορά των χρηματοδοτικών πόρων και αυτό θα είναι πραγματικά καταστροφικό. Mhm, δεν ξέρω αν απάντησα σε όλα. Μάλιστα. Σας ικανοποίησε η απάντηση. Ε, ναι. Με ικανοποίησε. Πράγματι, όμως το δεύτερο τμήμα του ερωτηματός μου μάλλον δεν απαντήθηκε που εντοπίζονται συγκεκριμένα τα εμπόδια, τα προσκόμματα. Είναι μια ομάδα χωρών, είναι ε, συγκεκριμένη πολιτική. Γιατί η Ευρώπη ενεργεί όπως ενεργεί. Υπάρχουν και αρνητικά παραδείγματα. Όμως πού μπορούμε να εντοπίσουμε τα εμπόδια που μας εμποδίζουν δηλαδή να φτάσουμε στην πράξη. Είναι τα Υπουργεία Μήνης. Γιατί εκείνοι λαμβάνουν τις ε, στρατητικές αποφάσεις. Σε ποιον λοιπόν θα πρέπει να απευθυνθούμε εμείς ως ευρωβουλευτές. Ε, Επιτρέψτε μου και εγώ να συμπληρώσω κάτι. Έχω την εντύπωση ότι και σε επίπεδο Υπουργείων Άμυνας αυτή η παλιά βρετανική σειρά, το Yes Minister, αυτό το σύριαλ πολλές φορές ε, είναι πράγματι αληθινό. Δηλαδή λαμβάνονται αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή Υπουργών Εξωτερικών. Μετά συναντιόνται άτυπα και Υπουργοί και όλοι συμφωνούν. Όμως ε, στο πλαίσιο των, ε, της διοίκησης είτε πρόκειται σε επίπεδο υπαλλήλων, είτε σε επίπεδο επιτελείων, των Υπουργείων, του Υπουργείου Άμυνα κυρίω, εκεί επικρατεί διαφορετική άποψη. Λένε yes, minister, ναι, ναι, κύριε Υπουργέ, αλλά πολλέ φορέ κάνουν ακριβώ το αντίθετο. Διότι σε διάφορε διαδικασίε ε, έχουν διασυνδέσει ε, με τη βιομηχανία, σχέσεις τις οποίες ε, καλλιεργούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ξαφνικά έρχεται ένας υπουργός με νέες τελείως διαφορετικές απόψεις και αυτό είναι ανήκουστο. Ως εκ τούτου έχω την εντύπωση ότι ανάμεσα στην ε, πολιτική ανακοίνωση και στην διοικητική εφαρμογή πολύ συχνά ε, παρεμβαίνουν εκείνοι που έχουν επιφυλάξει σε ε, στα αγγλικά σου να λέγαμε concern carriers, δεν ξέρω καν αν αυτό λέγεται στα αγγλικά, τέλο πάντων, λέει ο πρόεδρος, όσοι λοιπόν έχουν επιφυλάξει, σε τελική ανάλυση τα καταφέρνουν ε, την πολιτική άποψη ενός ε, υπουργού, ενός συμβουλίου ή ενός θεσμού να την αντιστρέψουν και πολλές φορές και να τη ματαιώσουν. Γι' αυτό λοιπόν όταν μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά ε, και πολλές φορές εδώ μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά με πολύ καλές ε, προθέσεις βέβαια θα πρέπει να προσέξουμε έτσι ώστε σε πολιτικό επίπεδο αυτοί που προϋπάρχουν και που τα ξέρουν όλα πολύ καλά να συμπεριλαμβάνονται και αυτοί στις διαδικασίες για να ε, προχωρήσει το όλο θέμα πολιτικά. Ίσως αυτό είναι λιγάκι άδικο και ίσως βέβαια ε, τα πράγματα να μην είναι έτσι ακριβώς σε όλες τις χώρες. Αλλά αν το λιγάκι στη Γερμανία το τι διαδραματίζεται και όπου πιστεύω ότι κάπως τα γνωρίζω τα θέματα, ξέρετε αυτή την εντύπωση έχω αποκομίσει, διότι ε, τις περισσότερες φορές συμφωνώ με την κυρία Υπουργό που έχουμε στη Γερμανία και εκεί δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πιο κάτω όμως ε, ως ε, Ευρωβουλευτής ε, εκεί δεν έχω πάρα πολλές επαφές και πολύ συχνά προκύπτει ότι σε ορισμένες διευθύνσεις δεν υπάρχει η απαραίτητη συνεργασία. Ίσως αυτό που σας έδωσα να είναι μια μερική απάντηση. Εγώ το διατύπωσα ως ερώτηση. Ο κύριος Μωρό είμαι σίγουρος ότι έχει εμπειρία και εκείνο από, από το πολιτικό και το δυτικό επίπεδο, το κατά πόσον συνεργάζονται ή αντιμάχονται η μία την άλλη πλευρά, θα μας πει ο ίδιο. Euh, Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να σας μεταφέρω την μαρτυρία μου ως προς αυτό. Να απαντήσω απευθεία στο ερώτημά σας. Υπάρχουν δύο ε, σημεία. Ένα στο οποίο δεν έχετε κάποια επιρροή και ένα άλλο στο οποίο έχετε. Που δεν έχετε τα κράτη-μέλη. Βρισκόμαστε σε μία κρίσιμη καμπή ή θα έλεγα ακόμα και ένα αδιέξοδο, όπου δεν μπορούμε να έχουμε ευρωπαϊκή άμυνα χωρίς τα κράτη-μέλη, γιατί εκείνοι έχουν τα οπλικά συστήματα, τη βιομηχανία, τις δυνάμεις, ε, την ε, εμπειρία και την ομοποίηση. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε να έχουμε ευρωπαϊκή άμυνα με τα κράτη-μέλη, επειδή δεν το επιθυμούν. Ούτε χωρίς λοιπόν, ούτε με τα κρατημέλη μπορούμε να την διαμορφώσουμε, γιατί δεν θέλουν, δεν επιθυμούν. Και όταν το λέω αυτό δεν εννοώ μόνο τις κυβερνήσεις, να το πούμε σαφώς. Έχουμε ευρωπαϊκά κρατημέλη που δεν επιθυμούν την ευρωπαϊκή άμυνα, γιατί θεωρούν ότι αυτή αντίκειται στα δικά τους συμφέροντα. Δεν θέλω να τους κατονομάσω, τους γνωρίζετε. Ε, μπορεί να προκαλέσει την αποχώρηση των Αμερικανών και το καθεξής. Υπάρχουν πολλά λοιπόν ευρωπαϊκά κρατημέλη που δεν επιθυμούν την ευρωπαϊκή άμυνα. Ακόμα όμως και μεταξύ αυτών που την επιθυμούν, την ευρωπαϊκή άμυνα, και μπορώ να φέρω και τη δική μου, όπως αναφέρω πέρα στη δική του, υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά μεταξύ του βαθέως κράτους, χωρίς να το αναφέρω συνωμοσιολογικά, όμως υπάρχουν διάφορα ε, επίπεδα και διοικητικά και βιομηχανικά και στρατητικά. Ε, υπάρχει λοιπόν μια διαφοροποίηση σχέση με αυτό που θέλουν ε, οι κυβερνήσεις. Σε μια μακιαβελική νότα λοιπόν, όταν αλλάζει η κατάσταση, δυσαρεστούμε αυτούς που έχουν επωφεληθεί από εκείνη και ακόμα δεν ευχαριστούμε αυτούς που θα ωφεληθούν. Είναι λοιπόν δύσκολη η μετάβαση από το ένα στο άλλο. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλοί που ε, είναι πολύ ικανοποιημένοι με την κατάσταση που έχει τώρα και στρατιωτικοί και βιομήχανοι και τα λοιπά. Ε, αν κάποιος ε, είναι ιδιαίτερα πλούσιος δεν χρειάζεται κάποια συνεργασία, γιατί να μπλέξει μέσα σε όλο αυτό εάν κάποιο έχει δυνατότητα να μη συνεργαστεί, δεν συνεργάζεται. Υπάρχει λοιπόν ένα, ε, ένας φυσικός φραγμός προς την συνεργασία. Εδώ λοιπόν δεν έχετε κάποια επιρροή στα κράτη-μέλη. Το δεύτερο εμπόδιο, στο οποίο έχετε όμως ε, αντίκτυπο, είναι ο τρόπος διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πάμε μπροστά όσο υπάρχει ομοφωνία. Αυτό να το ξέρουμε. Όλα τα υπόλοιπα είναι ε, φλιαρίες. Είδαμε και με τον ε, πρόεδρο Γιούγκερ, με, την, ε, με τη σύνοδο του Μέζελμπερικ μεταξύ Γαλλίας-Γερμανίας, υπέρ ενός ε, Συμβουλίου Ασφαλείας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δεν θα τα καταφέρουμε μεταξύ μα. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό το πρόβλημα πρώτα, γιατί εσύ, εσείς μπορείτε, μπορεί να μην καταφέρετε να κάνετε έναν αμυντικό σχεδιασμό ε, με 27 και 28 κράτη-μέλη μέσω τη ομοφωνία. Είτε θα μείνετε στους 27 και θα πάτε με την ειδική πλειοψηφία, είτε θα έχετε μια πρωτοπορία και θα βγείτε από το πλαίσιο των ε, ε, του καταστημένου όσο έχει τώρα. Όλα τα υπόλοιπα είναι λόγια. Okay. Λοιπόν, ε, αν ε, δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις ε, και αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την παρουσίαση της μελέτης και βεβαίως όλα αυτά που μας είπατε θα τα λάβουμε υπόψη. Όσον αφορά στις ε, περαιτέρω εξελίξεις, ε, θα παραμείνουμε σε επαφή. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, συστηματικά αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και τις προωθούμε. Ως εκ τούτου εμείς παραμένουμε δεσμευμένοι στην όλη υπόθεση. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά και όπως σας είπα θα παραμείνουμε σε επαφή. ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έκλεισε αυτό το θέμα της σημερινής διάταξης. Και πάμε τώρα με το σημείο υπαρθμών 12. Πρόκειται για το δεύτερο κύμα συνεργασίας με την διαρθρωμένη συνεργασία και θα ήθελα να έρθουν στο βήμα όσοι πρόκειται να λάβουν το λόγο.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 Attenzione tedesco. So. Eh, <laughs> so, eh. Λοιπόν, πάμε στο σημείο υπαριθμών 12. Το θέμα είναι το δεύτερο κύμα προγραμμάτων στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας ε, και θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά για άλλη μια φορά τον κύριο Αρναουτ Μόλινα, ο οποίος είναι ασκόν ε, διευθυντής χρέη διευθυντού, στο CMPD, ε, στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τον Λάρσα Σούμαν, ο οποίος ε, ασχολείται με θέματα ανάπτυξης ε, και ικανοτήτων στο στρατιωτικό επιτελείο και Αλεσάνδρο Τσινιόνι, ο οποίος είναι ο διευθυντής ε, της, ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Βεβαίως, ε, πριν από ένα χρόνο, χαρήκαμε που επιτέλους η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, η ΠΕΣΚΟ, ενεργοποιήθηκε και τις ε, οδηγίες ε, και το πλαίσιο για τις εργασίες της ΠΕΣΚΟ, αυτά τα λάβαμε υπόψη μας. Ήδη υπάρχουν ε, κάποια προγράμματα της ΠΕΣΚΟ, τα οποία τα έχουμε συζητήσει με παλαιότερες ευκαιρίες και θεωρούμε ότι κατ' ουσίαν βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο στο σωστό δρόμο να ενισχύσουμε την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρότι εγώ θέλω να επισημάνω ότι ορισμένα από τα προγράμματα, κατά την άποψη τη δική μου τουλάχιστον, θα έπρεπε να είναι λίγο πιο φιλόδοξα. Αυτό όμως είναι η δική μου προσωπική άποψη. Θα ήθελα να καλωσορίσω και τους τρεις ομιλητές, οι οποίοι θα μας εξηγήσουν αυτό το δεύτερο κύμα των ε, προγραμμάτων της ΠΕΣΚΟ. Θέλετε να ξεκινήσετε εσείς, παρακαλώ. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να πω ε, κάποια εισαγωγικά λόγια και μετά βέβαια οι συνάδελφοι από τα στρατιωτικά επιτελεία θα συμπληρώσουν. Να σας πω αυτής εξ αρχής ότι και οι τρεις μας ε, συνεργαζόμαστε εμείς προσωπικά αλλά και οι οργανισμοί τους οποίους εκπροσωπούμε για να στηρίξουμε την ΠΕΣΚΟ. Όσον αφορά τώρα το δεύτερο κύμα προγραμμάτων της ΠΕΣΚΟ, ας κάνουμε ένα βήμα προς τα πίσω και ας προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε ε, ποια είναι τα βήματα και διαδικασίες που εφαρμόζουμε ε, και οδήγησαν εχθές την απόφαση των Υπουργών να εγκριθούν τα επόμενα προγράμματα η απόφαση του Συμβουλίου, αυτή είναι η βασική απόφαση την οποία βασιζόμαστε, όπου προβλέφτηκε η ΠΕΣΚΟ και όπου προβλέφτηκαν συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Νομίζω είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι τα προγράμματα της ΠΕΣΚΟ είναι ένας τρόπος με τον οποίο τα κράτη-μέλη μπορούν να βοηθήσουν ε, να υλοποιηθούν οι υποσχέσεις τις οποίες ε, έχουν αναλάβει ε, μέσα από τη σύσταση της ΠΕΣΚΟ. Πρέπει λοιπόν, αυτό είναι το σχέδιο, να ε, εφαρμόσουμε αυτά τα προγράμματα και σε συνδυασμό με άλλες διαδικασίες. Όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, ακούσαμε με παλαιότερες ευκαιρίες ε, ε, τις απόψεις των κρατών μελών και γι' αυτό λοιπόν εμείς εμφανιζόμαστε ως το μόνο σημείο επαφής. Όσον αφορά στα προγράμματα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε πολλά και διαφορετικά προγράμματα. Ορισμένα ασχολούνται με την διαλειτουργικότητα, άλλα πάλι με το να προκύψουν νέες ικανότητες και υπάρχουν και προγράμματα που βασίζονται στη βελτίωση της επιχειρησιακής ε, εφαρμογής ε, των ικανοτήτων. Ε, τα κράτη-μέλη έχουν λάβει διάφορα προγράμματα. Υπάρχει ένας συντονιστής, ο οποίος κάνει και το συντονισμό. Τον Ιούνιο το Συμβούλιο ενέκρινε μία σειρά κανόνων ε, και αρχών για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται αυτά τα προγράμματα. Εδώ το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι όλα αυτά εντάσσονται στο ενωσιακό πλαίσιο ε, υπάρχουν δηλαδή οι διαδικασίες ε, που προβλέπουν την ε, ε, διασύνδεση ανάμεσα στα προγράμματα και το Συμβούλιο. Η διαδικασία για την επιλογή των προγραμμάτων, αυτή η διαδικασία ακολουθεί μία σειρά βημάτων. Πρώτον ως γραμματεία και μετά θα επεκταθούν οι συνάδελφοι. Έχουμε καθορίσει κριτήρια αξιολόγησης. Μετά ε, δημοσιεύουμε, προκυρήσουμε ένα διαγωνισμό έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να προτείνουν νέα προγράμματα. Αυτά τα προγράμματα τα αξιολογούμε εμείς η γραμματεία της ΠΕΣΚΟ από πλευράς ικανοτήτων ε, και κυρίως από το περισσότερο επιχειρησιακό πρίσμα. Και τέλος, η γραμματεία της ΕΠΕΣΚΟ είναι εκείνη η οποία κάνει τις τελικές συστάσεις και οι οποίες μετά από σύσταση ε, της προσώπου ε, μεταβιβάζονται στο Συμβούλιο. Αυτά γίνονται αρχές Οκτωβρίου. Ε, κατ' ουσίαν τώρα το όλο θέμα είναι στο Συμβούλιο και η στρατιωτική επιτροπή έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και έτσι λοιπόν έχει δημιουργηθεί βάση για την απόφαση του Συμβουλίου, η απόφαση η οποία λήφθη εχθές. Ε, τα προγράμματα κατά τη δική μας άποψη είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Είναι νέα προγράμματα τα οποία μεταξύ άλλων έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν τα κενά που έχουν εντοπιστεί σε σχέση με τις αναληφθήσεις δεσμεύσει. Η φιλοδοξία μας είναι να ενισχύσουμε τις ικανότητές μας, να υπάρχει διασύνδεση, ε, να αναπτύσσουμε τις δυνάμεις μας ε, και επίσης να συνεργαστούμε όλο και περισσότερο για να αντιμετωπίζουμε τις απειλές που ε, αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις μας στα, στα θέατρα των επιχειρήσεων. Όσον αφορά λοιπόν αυτά τα προγράμματα της ΠΕΣΚΟ, σα είπα, αυτές λήφθη απόφαση σε επίπεδο συμβουλίου. Ε, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι υπάρχει και μία νέα ιστοσελίδα της ΠΕΣΚΟ, η οποία από τις 5 σήμερα το απόγευμα θα δημοσιευτεί και εκεί θα διατίθενται από την ΠΕΣΚΟ όλες οι απαραίτητες πληροφορίες στο κοινό, στην κοινή γνώμη. Εχθές η συζήτηση στους υπουργού κατέδειξε τη σημασία όχι μόνο αυτών των νέων προγραμμάτων, εχθές ε, οι υπουργοί εστιάστηκαν και στην εφαρμογή. Του χρόνου έχουμε το καθήκον να εξετάσουμε τα ε, συμπεράσματα που μπορούμε να εξάγουμε από τη διαδικασία που ακολουθήθηκε εφέτος, έτσι ώστε να προκύψει ο νέος ετήσιος κύκλος για την επόμενη χρονιά. Οφείλουμε λοιπόν να αναφερθούμε στο Συμβούλιο για την πρόοδο που θα έχει επιτευχθεί μέχρι την Άνοιξη. Και με αυτά θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλό απόγευμα σε όλους. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε ως μέλος της γραμματείας της ΠΕΣΚΟ. Από επιχειρησιακή άποψη θα ήθελα να σα εξηγήσω με περισσότερες λεπτομέρειες πώς ακριβώς κάναμε την αξιολόγηση λοιπόν από επιχειρησιακής άποψη. Ο κύριος Μόλεναρ ήδη ανέφερε ότι τα έργα ΠΕΣΚΟ θα πρέπει να αποτελέσουν και ένα, ένα όχημα πλήρωση ε, πλήρωσης των δεσμεύσεων και εμείς Έχουμε εξετάσει ιδίω τη δέσμευση 12 που έχει να κάνει με την διαθεσιμότητα και δυνατότητα ανάπτυξη δυνάμεων και ικανοτήτων. Εξετάσαμε την δέσμευση 13 που έχει να κάνει με τη διαλειτουργικότητα των δυνάμεων που είναι πολύ σημαντική από επιχειρησιακή άποψη, καθώ και τι δεσμεύσει που άπτονται των ε, ελλείψεων ικανότητας. γιατί οι προϋποθέσεις ε, τίθενται πίσω από την UAMS. Και τέλος, εξετάσαμε και τη δέσμευση 10, που έχει να κάνει με την κοινή χρήση υφιστάμενων δυνάμεων, που δηλαδή υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης των υφιστάμενων δυνάμεων για να διαμορφώσουμε ένα σύνολο δυνάμεων που μπορεί να αναπτυχθεί σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αυτά εξετάσαμε από πλευρά δεσμεύσεων. Μετά έχουμε και αναπτύξαμε ειδικά κριτήρια αξιολόγησης που συνοδεύουν τα όσα σας προανέφερα. Πρώτον, η ευθυγράμμιση με τον κατάλογο ε, απαιτήσεων και προποθέσεων του 2017. Ποιες είναι δηλαδή οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από συγκεκριμένα σενάρια, που είναι ρεαλιστικά και εύλογα από πλευράς σχεδιασμού. Δεύτερον, εξετάσουμε τον κατάλογο προόδου. Απαιτήσει δηλαδή που αυτή τη στιγμή δεν πληρούνται από τα κράτη-μέλη, που υπάρχουν ελλείψεις και δυναμίες. Τρίτον, η ευθυγράμμιση με διδάγματα του παρελθόντος από τις επιχειρήσεις. Τι είδους διδάγματα έχουμε αντλήσει, πού έχουμε εντοπίσει κενά στις επιχειρήσεις μας. Μετά, τέταρτον. Δυνατότητα αξιοποίησης των δυνάμεων και κατά πόσο είναι πιθανόν οι δυνάμεις που θα προκύψουν από ένα έργο να αναπτυχθούν ε, σε μία στρατιωτική επιχείρηση. Employability και deployability. Μετά, εξετάσαμε πού και κατά πόσο οι ικανότητες συμβάλλουν στην βελτίωση της διαλειτουργικότητας των δυνάμεων. Ιδίως όταν έχουμε να κάνουμε με πολυεθνικές δυνάμεις η διαλειτουργικότητα δεν είναι δεδομένη. Και γι' αυτό προσπαθήσαμε να βρούμε συγκεκριμένα έργα που ενισχύουν τη διαλειτουργικότητα. Τέλος, διαθεσιμότητα δυνάμεων. Παρότι η διαθεσιμότητα εξαρτάται και από τη βούληση και την προθυμία των πρώτων μελών να διαθέσουν τις δυνάμεις. Επομένω, ε, περισσότερο μαντεύουμε παρά γνωρίζουμε. Εξετάσαμε όλες ε, τις ε, προτάσεις έργου, 33 υπευλήθησαν από τα κράτη-μέλη. Είχαμε 6 εβδομάδες και συμπεριλάβαμε όλα τα πεδία ενδιαφέροντος, όλες τις διευθύνσεις χρησιμοποιήσαμε όλη τη διαθέσιμη εμπειρογνωμοσύνη. Από επιχειρησιακής άποψης, αυτές οι προτάσεις που θεωρήθηκαν πιθανές, πιθανά έργα ΠΕΣΚΟ και ε, τα επιλέξαμε χθε έχουν να κάνουν με τη βελτίωση της ε, βράχη και μακροπρόθεσμης ικανότητας και αποτελεσματικότητας σε στρατηγικό επίπεδο. Και υπογραμμίζουμε ότι ε, συνεχίζουμε και ακολουθούμε τη δυναμική ΠΕΣΚΟ και θέλουμε να πετύχουμε τα αποτελέσματα, όμως θέλουμε να εντοπίσουμε και συνέργειες μεταξύ ΠΕΣΚΟ και αυτού που ανέφερε ο Πρόεδρος προηγουμένως, ότι το ΚΑΔ έχει και στηρίζει την ανάπτυξη ικανοτήτων και γι' αυτό είναι σημαντικό να ε, συνδέσουμε τα ευρήματα CAD με την ΠΕΣΚΟ και την επιλογή έργων στο πλαίσιο ΠΕΣΚΟ. Τέλος, να πω ότι πρέπει να δούμε συνολικά την ΠΕΣΚΟ και όχι επιμέρους έργα ΠΕΣΚΟ. Δεν πρέπει λοιπόν να ξεχνάμε τη συνοχή μεταξύ των έργων ΠΕΣΚΟ. Θα σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα. Από τα 17 νέα έργα επιλέγω ένα. Ένα πακέτο ικανότητας ε, υποβρύχιων παρεμβάσεων που θα λαμβάνει υπόψη ε, πολλούς διαφορετικούς εξοπλισμούς, ε, υποβρύχιους ή και υποβρύχια μη επανδρομένα σκάφη και διάφορα άλλα στοιχεία. Έχει λοιπόν να κάνει με υλικό, με εξοπλισμό, με κατάρτιση, εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι από μόνο του αυτό το έργο καλύπτει πάνω από μία πτυχή της ικανότητας. και θα συνδεθεί και με άλλα έργα ΠΕΣΚΟ που ήδη έχουν ξεκινήσει, όπως η προστασία λιμένων ή και το MCM, το σύστημα MCM. Παρότι λοιπόν εκ πρώτης όψεως αυτή η πρόταση φαίνεται να μην προσφέρει πολλά, απλώς μια σχολή κατάδυση ας πούμε. Ε, αν το δείτε συνολικά σε πλαίσιο, στο πλαίσιο ΠΕΣΚΟ, η αξία που επιφέρει είναι πολύ μεγαλύτερη. Και αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα κατά νου. Κατά την αξιολόγηση έργων. Δεν είναι μόνο το κάθε επιμέρους έργο που πρέπει να εξετάζουμε, αλλά συνολικά η συνεκτική εικόνα του πακέτου. Και θα μείνω εδώ. Κύριε Τσινιώνη, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ ε, και τους ακρατές που είναι εδώ σήμερα. Θα είμαι σύντομος. Θέλω απλώ να ευκρινίσω και να συμπληρώσω τα όσα είπα προηγούμενοι μιλητέ. Ανέφερε ο κύριο Μόλεναρ την, ε, την ευρύτερη διαδικασία για την υποβολή σχεδίων ΠΕΣΚΟ και την επιλογή των έργων. Ε, ο προηγούμενο ομιλητή, ε, κύριο Σούμαν, παρουσίασε τα κριτήρια αξιολόγηση αυτών των έργων από επιχειρησιακή άποψη. Και εγώ θα σα πω δύο λόγια παραπάνω για τα κριτήρια που χρησιμοποιήσαμε για την αξιολόγηση των προτάσεων έργου που έφτασαν στην γραμματεία της ΠΕΣΚΟ από πλευράς ικανότητας. Δώσαμε λοιπόν στα κράτη-μέλη ορισμένα στοιχεία για να λάβουν, ε, να είναι σε καλύτερη θέση να πάρουν αποφάσεις σε ό,τι αφορά την επιλογή ε, project στο πλαίσιο ΠΕΣΚΟ. Από πλευράς ικανοτήτων λοιπόν εξετάσαμε πράγματα από μέσο και μακροπρόθεσμη προσέγγιση. Για να δούμε πώς αυτά τα έργα διαμορφώνουν το μέλλον της συνοχής ε, των ευρωπαϊκών δυνάμεων και ικανοτήτων. Πώς το κάναμε αυτό. Προσπαθήσαμε να απαντήσουμε σε τέσσερις βασικές ερωτήσεις. Πρώτον, κατά πόσο το έργο θα συμβάλλει στη βελτίωση της συνοχής ε, των ευρωπαϊκών ικανοτήτων. Εντάξει, αρκετά αφηρημένο ερώτημα. Εξετάσαμε τις συμπεφωνημένες προτεραιότητες ικανοτήτων των κρατών μελών, που συμφώνησαν δηλαδή να ακολουθήσουν τα κατημέλη για την ανάπτυξη ικανοτήτων. Και αναφέρθηκε προηγουμένως και το CAD, που είναι μια συντονισμένη αιτήσια αναθεώρηση για την άμυνα. Εξετάσαμε και τα αποτελέσματα αυτής λοιπόν για να δούμε κατά πόσο αυτά τα δύο συμβαδίζουν. Και μετά προσπαθήσαμε να δούμε τον αντίκτυπο του κάθε έργου στο ευρύτερο πλαίσιο. Βέβαια, πρέπει να δούμε αν πρόκειται για ένα θαλάσσιο έργο, πρέπει να δούμε τι γίνεται στον θαλάσσιο τομέα. Και ποια θα είναι η επίδραση αυτού του έργου μέσω και μακροπρόθεσμα. Ένα άλλο στοιχείο είναι η οριμότητα του έργου. Ξετάσαμε τις ε, προϋποθέσεις. Όταν έχουμε να κάνουμε με συνεργασία με πολλά κράτη-μέλη, πρέπει να καταλήξουμε σε κοινέ ε, προδιαγραφές. Κάποια έργα λοιπόν μπορεί να είναι πιο όρημα και να βασίζονται σε υφιστάμενες κοινέ προδιαγραφές, αλλά προσπαθούν να τις αναπτύξουν. Άλλο σημαντικό στοιχείο που έχει να κάνει με την οριμότητα είναι η συνοχή με ήδη φυστάμενες και συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Υπάρχουν περιφερειακές δραστηριότητες για την ανάπτυξη ικανοτήτων ή μπορεί να πρόκειται για έναν άλλο τομέα, αλλά να άπτεται κάπως της ευρωπαϊκής ικανότητας. Πρέπει να τα δούμε λοιπόν σφαιρικά για να δούμε αν υπάρχουν συνέργειες, αν υπάρχει συνοχή, δεν πρέπει να υπάρχουν άλλοι επικαλύψεις. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Μετά, εξετάζουμε και τη συνοχή στο πλαίσιο των ε, προσπαθειών ε, στον άτομο, την κοινή διακήρυξη. Και εκεί λοιπόν εξετάζουμε την ε, συνοχή με άλλες νατοικές ενέργειες και κατά πόσο ένα έργο πληρεί και ορισμένες ε, προτεραιότητες του ΝΑΤΟ. Τέλος, εξετάζουμε και την οικονομική και βιομηχανική διάσταση. Βέβαια, το πιο σημαντικό είναι το πρώτο. Από πλευράς ικανοτήτων, λοιπόν, το πιο σημαντικό είναι αν κάπως συνδέεται με την αύξηση ικανοτήτων ε, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Έχουμε 34 έργα αυτή τη στιγμή. Η καλύτερη προσέγγιση είναι να τα εξετάζουμε από κοινού και ανάλογα με τον τομέα. Κάποια συμβάλλουν ε, στην ε, κατάρτιση, στην εκπαίδευση, στη διαμόρφωση κοινών ε, μηχανισμών διευκολύνσεων εγκαταστάσεων. Άλλα επικεντρώνονται στο χερσαίο σκέλος, άλλα στο θαλάσσιο τομέα. για τη στήριξη της συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα. Μετά στον εναέριο τομέα υπάρχει μια ομάδα έργων που ε, συμβάλλουν στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και σε ό,τι έχει να κάνει με το συγκεκριμένο σύστημα, το πληροφορικό σύστημα και σύστημα επικοινωνιών. Και εγκάρσια έργα που θα μας δώσουν ικανότητες που θα αξιοποιήσουμε σε διάφορους τομείς και τέλος έχουμε συγκεκριμένο έργο ε, που έχει να κάνει με το διάστημα και αυτό πολύ σημαντικό στο πλαίσιο ΠΕΣΚΟ και θα μείνω εδώ Πρόεδρε Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνάλφοι, τώρα έχουν το λόγο. Κυρία Λούζινγκ. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου ευθύ εξ αρχή να πω το εξή. Θα το έβρισκα πάρα πολύ καλό να έχουμε ένα κατάλογο αυτών των ε, προγραμμάτων. Βέβαια, αυτά συμβαίνουν σε μια τέτοια χρονική στιγμή όπου ε, κατ' ουσίαν λαμβάνονται αποφάσει στο Συμβούλιο. Δεν πιστεύετε λοιπόν ότι θα ήταν σκόπιμο ε, να ασχοληθούμε και εμείς με το θέμα αυτό σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, αλλά αυτό να έχει ήδη λάβει χώρα, να έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Αυτή προφανώς και είναι μια καθαρά ρητορική πολιτική ερώτηση. Τώρα, θα ήθελα περισσότερο με λεπτομέρειες να απευθυνθώ στους ομιλητές και να ρωτήσω το εξή. Από ό,τι φαίνεται, ο κατάλογος αυτός περιείχε αρχικά 33 προτάσεις και τελικά απέμειναν 15. Ποια ακριβώς προγράμματα διαγράφηκαν και για ποιο λόγο. Όσον αφορά αυτό τον κατάλογο των προγραμμάτων, δεν είδα να αναφέρεται και το κόστος. Ως εκ τούτου, ε, ποιο είναι το κόστος και το χρονικό διάστημα που προβλέπετε. Ας πάρουμε ως παράδειγμα τα Eurodrones. Δηλαδή, γι' αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα έχετε υπολογισμό κόστους και χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άλλες ερωτήσεις, η κυρία Βαλέρο. Θα ήθελα να ε, κάνω μια ερώτηση και συγκεκριμένα και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω για τα drones. Ορισμένοι στο Κοινοβούλιο επιθυμούν να υπάρχει μια ε, κοινή στάση επ' αυτού του θέματος. Να υπάρχει κοινή στάση από το Συμβούλιο όσον αφορά το ενδεχόμενο χρήση των drones. Μήπως μπορείτε να τοποθετηθείτε παρακαλώ επ' αυτού. Και εμείς, και εγώ ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ε, και θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιες συμπληρωματικέ ερωτήσεις και οι δύο συνάδελφοι έθιξαν τα drones. Είναι το πιο γνωστό πρόγραμμα και γι' το λόγο το θίγουμε όλοι. Ε, θέλω να σας πω, χαίρομαι ιδιαίτερα ε, που ε, υπάρχει αυτό το πρόγραμμα το οποίο και ως πρόγραμμα της ΠΕΣΚΟ μπορεί λιγάκι να ξεφύγει από το δικό μας το πρόγραμμα και να υποφεληθεί. Έτσι, μία πιο γενική ερώτηση και με βάση αυτά που ελέγχθησαν στο προηγούμενο σημείο της μέσης διάταξη από τον συνάδελφό μας, να πω το εξής. Υπάρχει το εξής ερώτημα. Αυτή τη φορά τα προγράμματα σε ποιο βαθμό προέκυψαν από στρατηγικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δηλαδή έχουμε ήδη ορίσει το τι θα επιθυμούσαμε να έχουμε ε, ως capabilities, ως ικανότητες. Ή μήπως πρόκειται έτσι ένα είδος συμβιβασμού εθνικά προγράμματα τα οποία ε, όλα ε, συνδυάστηκαν. Πού είναι τελικά αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα που ακολουθούν μια ευρωπαϊκή στρατηγική και έχουν ως στόχο να κλείσουν κενά. Πράγματι τα Eurodrones είναι ένα κλασικό πρόγραμμα όπου ισχύει κάτι τέτοιο. Και κάτι άλλο. Έχουμε και το ε, πρωτόκολλο 10 το οποίο αφορά ε, στις κοινέ μόνιμες ε, ενώσεις, οι επιτροπές. Πού βρίσκονται αυτές, δεν τις βλέπω, δεν υπάρχουν. η συμμετοχή σε εθνικές, ε, μάλλον σε υπερεθνικές ένοπλες δυνάμεις, αυτή η συμμετοχή δεν προβλέπεται πουθενά στα προγράμματα. Και τελικά, μήπως είναι μόνο εθνική κατάλογη. Αν δούμε το πρόγραμμα ε, European High Atmosphere Platform, νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα απλά και μόνο το συμπεριλάβαμε, το επιθυμούσαν οι Γάλλοι, γιατί το έχουν ήδη οι Αμερικανοί. Ε, αυτός είναι ο λόγος ή μήπως πράγματι υπήρχε μια ευρωπαϊκή ανάγκη η οποία εντοπίστηκε. Σας το λέω έτσι αυτό ενδεικτικά για να μας πείτε κατά πόσον ο κατάλογος αυτός είναι τελικά ευρωπαϊκός ή είναι απλά η σύνθεση των εθνικών επιθυμιών. Δεν ξέρω, υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Παρακαλώ. Σας ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ε, νομίζω ότι η Ιρλανδία δεν συμμετέχει σε κανένα από τα νέα προγράμματα. Αναφερθήκατε στην έστω σελίδα της ε, την νέα ιστοσελίδα της Πέσκο, μπορείτε να μας την πείτε ποια είναι, για να μπορούμε να μπούμε, να τη δούμε λιγάκι την ιστοσελίδα αυτή. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Yeah, okay. I, I will start, uh, with Θα ξεκινήσω απαντώντας στο πρώτο ερώτημα. Για τις προτάσεις που λάβαμε πώς φτάσαμε στα 17 και με ποια διαδικασία. Όλες οι προτάσεις που υποβλήθηκαν ήταν πολύ σημαντικές. Ήταν σημαντικές και για τα κράτη-μέλη. Έργα που μας ενδιέφεραν. Πολύ σημαντικά. Όμως ως γραμματεία ΠΕΣΚΟ μαζί με τα κράτη-μέλη συμφωνήσαμε να χρησιμοποιήσουμε σειρά κριτηρίων για να εξετάσουμε κάθε πρόταση ξεχωριστά και να ενημερώσουμε καλύτερα τα κράτη-μέλη. Πώς, ε, κατά πώς ανταποκρίνονται οι προτάσεις με τα κριτήρια που καθορίσαμε. Επομένως, ο συνάδελφος Σούμαν και εγώ περιγράψαμε τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων Εξετάσαμε κάθε πρόταση λοιπόν για έργο με βάση όλες τις προοπτικές, με βάση όλες τις οπτικές γωνίες. Κάναμε διασταυρούμενη ανάλυση ικανοτήτων και επιχειρησιακής ετοιμότητας, capability και operation και καταλήξαμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και τελικά καταλήξαμε σε 17 project που τα διάλεξαν τα κράτη-μέλη. Όσο ε, Γενική Γραμματεία κάναμε αμερόληπτη αξιολόγηση με βάση αυτά τα κριτήρια και αυτές τις οπτικές γωνίες capability και operation και δώσαμε την αξιολόγηση στα κράτη-μέλη. Και τα κράτη-μέλη μετά διάλεξαν ποιο ήθελαν να εφαρμοστεί στο πλαίσιο ΠΕΣΚΟ. Αυτή ήταν η διαδικασία και έτσι φτάσαμε στον κατάλογο των 17 που σας ανακοινώσαμε. που ανακοίνωσε το Συμβούλιο. Για το Eurodrone μιλούμε για ένα έργο που χτίζεται πάνω σε ένα άλλο έργο που ήδη υπάρχει και που είναι αρκετά όριμο Medium Altitude Long Endurance Type System. Σύστημα δηλαδή μέσης αντοχής υψηλού υψομέτρου για ε, δράσεις εποπτείας και αναγνώρισης. Αυτά. Και μετά να απαντήσω και στο τελευταίο. No, Ευχαριστώ και εγώ, λέει ο κύριος Μόλεναρ. Μέρος της αξιολόγησης είναι να εξετάζουμε τα project. Εάν τελικά δεν βρίσκονται στο τελικό κατάλογο, ναι, δεν εξαφανίζονται. Μπορούν τα κράτη-μέλη να υποβάλουν βελτιώσεις και να τα ξαναπροτείνουν. Η τεχνική αξιολόγηση δεν ήταν θετική για εμάς. Τώρα για το κόστος και για τον προϋπολογισμό των διαφόρων project αυτό είναι στα χέρια των κρατών μελών. Δεν υπάρχει κοινό προϋπολογισμός. Εμείς από τεχνική σκοπιάς, και αυτό είναι μέρος της οριμότητα ενό έργου, εξετάζουμε κατά πόσο υπάρχει διεθνικό σχεδιασμός χρηματοδότησης, εάν υπάρχει σχέδιο να διατεθούν αυτά τα κονδύλια. Γιατί στην τελική αυτό είναι και ο μόνο τρόπο για να ε, ευοδοθεί αυτό το έργο. Αλλά δεν ελέγχουμε το κόστος αυτό καθεαυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο πώς λειτουργεί τελικά, είναι μια προσέγγιση bottom-up, από κάτω προς τα πάνω. Οι συμμετέχοντες, τα κράτη-μέλη υποβάλλουν προτάσεις, συνεργάζονται με τα κράτη-μέλη συμμετέχοντες για να τα ειδοποιήσουν και εμείς κάνουμε top-down αξιολόγηση, από πάνω προς τα κάτω αξιολόγηση. Κατά πόσο αυτά που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρούνται οι προδιαγραφές και ούτω καθεξής. Άρα, για την ενσωμάτωση των έργων δουλεύουμε από κάτω προς τα πάνω και για την αξιολόγηση αυτών δουλεύουμε από πάνω προς τα κάτω. Τώρα, μπορούμε να πάμε ακόμα πιο πέρα. Δεν μπορούμε όμως ακόμα να πούμε από ψηλά εμείς άνωθεν, κοιτάξτε εσείς εκεί κάτω κάντε ένα έργο για το χύψη θέμα. Αυτό δεν είμαστε έτοιμοι να το πούμε κατώ, ακόμα. Ίσως τα κράτη-μέλη που κάνουν το δικό τους σχεδιασμό, που βάζουν και τα δικά τους κονδύλια. Ενδιαφέρον είναι ο σύνδεσμος μεταξύ των έργων που γίνονται για το EDPIP, κάποια έργα ΠΕΣΚΟ που ε, παρουσιάζουν ενδιαφέρον μπορεί να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση βάσει και αυτού του εργαλείου. Τώρα, για την Ιρλανδία και για άλλες χώρες που δεν έχουν συμμετάσχει σε έργα. Σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι είναι μεγάλο το ενδιαφέρον των κρατών μελών, μεγάλο το βάρος, αλλά είναι και δαπανηρό, χρειάζεται χρόνο και επένδυση μεγάλη. Δεν με εκπλήσει λοιπόν κάποια κράτη-μέρη να καταλήξουν όχι για πολιτικούς λόγους αλλά για λόγους δυνατοτήτων ότι απλά δεν δίνανται. Δεν είναι αυτό μέρος των δυνατοτήτων τους. pesco.europa.eu Αυτή είναι η νέα ιστοσελίδα. Και όλα αυτά ε, έγιναν και με τη βοήθεια των συναδέλφων από το EDPA. Και εγώ θα ήθελα κάτι να προτείνω. για τις συνολικές στρατηγικές πώς ταιριάζουν στη συνολική διαδικασία. Το CDP, Capability Development Plan, καθοδηγείται από τη συνολική στρατηγική και το εφαρμοστικό σχέδιο. και τα διάφορα σενάρια τα οποία προκύπτουν από αυτή την συνολική στρατηγική, την Global Strategy. Άρα, ό,τι ζητούμε ως capabilities, ως ε, δυνατότητες, προκύπτει από την αποστολή, από τις ε, δράσεις, από τη συνολική στρατηγική. Άρα, όποια απέτηση και αν έχουμε, τελικά προκύπτει από τα στρατηγικά μας έγγραφα. Και για εμάς αυτό είναι το πιο σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης. Και υπάρχουν και μειονεκτήματα. Επομένως, για μένα, είναι σαφής η σύνδεση με τις συνολικές στρατηγικές. Ευχαριστούμε. Να δώσω πάλι το λόγο στην κυρία Λόιζινγκ. Μετά Βαλέρο και Φλάναγκαν, παρακαλώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για ένα πλαίσιο δράσης πραγματικά καινοτόμο. Είναι κάτι το απολύτως καινούριο. Και εμείς, ε, τρόπον την Α, είμαστε το ελεγκτικό όργανο, το κοινοβουλευτικό. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ρωτήσω το εξή. Όσον αφορά αυτό το πρόγραμμα με τα drones υπάρχει και το θέμα του χρονοδιαγράμματος. Δηλαδή θα ήθελα να γνωρίζω κατά πόσον έχετε περισσότερες λεπτομέρειες από αυτού του προγράμματος. Είπατε ότι δεν έχετε λεπτομερή αναφορά του κόστους, αλλά παρόλα αυτά μήπως έτσι μπορείτε να μας αναφέρετε μια τάξη μεγέθους σχετικά με το κόστος. Γιατί νομίζω είναι σημαντικό οι πολίτες των κρατών μελών να έχουν έτσι μια ιδέα πόσο θα κοστίσει όλο αυτό. Και κάτι άλλο, δεν απαντήθηκε ένα άλλο δικό μου ερώτημα. Δηλαδή, εγώ δεν σας ρώτησα τόσο για τη διαδικασία, πώς ε, δηλαδή απορρίπτονται τα προγράμματα, αλλά να μας αναφέρετε παραδείγματα πώς ακριβώς ε, απορρίπτονται. Ε, υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα. Ποια είναι τα προγράμματα που απορρίφθηκαν. Και επειδή εσείς ο ίδιος είπατε ότι έχετε καθορίσει κάποια κριτήρια για την απόρριψη, ποια ακριβώς είναι αυτά τα κριτήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η συνάδελφος κυρία Βαλέρο. Και εγώ σε σχέση με το αρχικό ερώτημα, κατά πόσο αυτά ταιριάζουν με το σχέδιο ανάπτυξης ικανοτήτων και Capability Development Plan. Είπατε ότι είναι μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω και όχι από πάνω προς τα κάτω. Πώς ταιριάζει αυτό με την ευρωπαϊκή αξιολόγηση που γίνεται από πάνω προς τα κάτω. Το CDP είναι κριτήριο για την αξιολόγηση, έτσι δεν είναι αυτό καταλάβα ότι είπατε για την αναγνώριση, για την έγκριση αυτού του έργου, έτσι δεν είναι. Ε, thank you, ε, Mr. Ευχαριστώ. Για την Ιρλανδία, ο κύριος Μόλεναρ απάντησε στο ερώτημα για το κατά πόσο υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν αποσυρθεί από αυτά τα έργα. Και όταν απαντούσατε, είπατε ότι ε, υπάρχουν χώρες που θεώρησαν ότι είναι beyond their capacity, πέρα από τις ε, δυνατότητές τους. Είμαστε πλούσια χώρα τώρα. Πιστεύετε ότι γι' αυτό το λόγο δεν συμμετείχαν. Ή τέλο πάντων κάποιοι δηλαδή έχουν χρήματα και έχουμε το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, όταν λέτε beyond their capacity, πέρα από τι δυνατότητέ του, δεν το λέτε με την οικονομική σκοπιά, αλλά με την έννοια των δεσμεύσεων, της υπευθυνότητα, της ανάληψης ευθύνης. Τι εννοείται ακριβώ όταν είπατε ότι κάποιε χώρε δεν συμμετείχαν γιατί ήταν πέραν από τι δυνατότητέ του και αποσύρθηκαν. Ποιο θέλει να απαντήσει. Ο κύριος Τσινιώνει. Ναι, θα προσπαθήσω να είμαι πιο συγκεκριμένος, να απαντήσω ίσως με το δεύτερο ερώτημα, να ξεκινήσω πρώτα, ε, που είναι πιο σύντομο. Για το CDP, τι προτεραιότητες και κατά πόσο είναι από πάνω προς τα κάτω ή από κάτω προς τα πάνω. Κοιτάξτε, οι προτεραιότητες για την ανάπτυξη ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι προτεραιότητες που έχουν προσδιορίσει τα κράτη-μέλη. Άρα, προσδιορίζουν σε ποιους τομείς έχουν προτεραιότητα και θέλουν να αναπτύξουν δυνατότητες με συνεργατικό τρόπο. Άρα κάποιες εθνικές προτεραιότητες ευθυγραμμίζονται με τις ευρωπαϊκές. Οι προτεραιότητες CDP προέρχονται από τέσσερις τομείς. Τα διδάγματα που έχουν αντληθεί, τις αποστολές που έχουν γίνει, τα μειονεκτήματα, τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί. Και άρα είχαμε μακροπρόθεσμη κάτοψη του ποια και capabilities θέλουμε να αναπτύξουμε, πού επενδύουν τα κράτη-μέλη και πού, σε ποια σημεία θέλουν να συνεργαστούν. Το θεωρώ φυσικό να υπάρχουν αυτές οι δύο διεργασίες. Τα κράτη-μέλη πρέπει να προβληματιστούν για το πώς θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις προτεραιότητες, πώς θα τις δρομολογήσουν. Κάθε project είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και από την ευρωπαϊκή οπτική γωνία και από πλευρά CDP είναι σημαντικό τα έργα να ε, αντιστοιχούν στις προτεραιότητες. Τώρα για τα κριτήρια. Τι είδους κριτήρια χρησιμοποιήσαμε. Ίσως ήμασταν υπερβολικά τεχνικοί στην ενημέρωση και σταθήκαμε πολύ σε τεχνικά σημεία. Να τονίσω όμως το εξής. Τα κριτήρια που ανέφερα στην ενημέρωση που σας έκανα. Το κριτήριο που χρησιμοποιούμε από πλευράς capability, δηλαδή να δούμε μεσομακροπρόθεσμα ε, πώς θα αναπτυχθεί αυτή, αυτό το capability, αυτό είναι και το βασικό μας κριτήριο. Άρα, όταν σας υπενθυμίζω τα τέσσερα βασικά ερωτήματα στα οποία προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις, αυτό ακριβώς το εγχείρημα, η απάντηση στα ερωτήματα και τα στοιχεία τα αποδεικτικά ε, που κομίζουν τα project, τα έργα, είναι τα βασικά κριτήρια για να τα δεχτούμε. Και στη δική του ενημέρωση Ο κύριος Σούμαν αναφέρθηκε στο στρατιωτικό σκέλος ότι οι στρατιωτικοί είναι αυτοί που εξέτασαν το επιχειρη... την επιχειρησιακή πτυχή. Με αυτά τα κριτήρια λοιπόν δώσαμε πληροφορίες στα κράτη-μέλη για να διαλέξουν τα έργα που θέλουν. Άρα δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο απόρριψη γιατί δεν απορρίψαμε κανένα project ως γραμματεία ΠΕΣΚΟ αλλά κάναμε αξιολόγηση των προτάσεων με βάση κριτήρια που είχαμε ανακοινώσει και είχαμε ε, δώσει στα κρατη και τα ήξεραν. Και με βάση αυτά τα κριτήρια ενημερώσαμε τα κράτη-μέλη. Άρα μιλούμε για capabilities, για ικανότητες που αναπτύσσουν τα κράτη-μέλη, εννοώντας ότι τα κράτη-μέλη είχαν ήδη την ευκαιρία, αλλά και τη δυνατότητα να αποφασίσουν τι ακριβώς θέλουν να αναπτύξουν στο πλαίσιο της ΠΕΣΚΟ. Γραμματιακά λειτουργήσαμε δηλαδή στηρίζοντας τα κράτη-μέλη. Uh, add... Να προσθέσω και το εξή λέει ο κύριος Σούμαν. Μας ρωτήσατε για τα έργα που δεν έχουν επιλεγεί. Και στράφηκα προς τον συνάδελφο, γιατί δεν έχω τον κατάλογο με τις 33 προτάσεις, ούτε εκείνος τον είχε, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να σας δώσω δύο παραδείγματα και να εξηγήσω γιατί τελικά δεν τα προτείναμε αυτά τα δύο έργα στα κράτη-μέλη για να επιλεγούν. Strategic Air Lift. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι δυνατότητες αερομεταφοράς εξοπλισμού σε μεγάλες αποστάσεις. Ε, ε, ε, έχουμε λήψεις, πάρα, πολλές, πάρα πολύ μεγάλες ελλείψεις. Αυτή η πρόταση θεωρήθηκε εξαιρετικά πολύτιμη. Δυστυχώς όμως, μόνο το, προ... το κράτος μέλος που το πρότεινε ήταν έτοιμο να ξεκινήσει μια τέτοια πρόταση την υλοποίησή της. Ούτε ένα άλλο κράτος μέλος δεν ήθελε και δεν μπορούσε να προσχωρήσει σε αυτό το έργο. Άρα, εάν ένα, ένα κράτος ε, μέλος το επιθυμεί και μπορεί να το πράξει, ε, αυτό δεν είναι ενωσιακό έργο. Δεύτερο παράδειγμα μία πρόταση για την, ε, το, προστατευτικό επίχρησμα είναι μια δική μπογιά του εξοπλισμού που το κάνει τον εξοπλισμό το υλικό λιγότερο εύκολα εντοπίσιμο από τα ραντάρ. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα τεχνική λύση, αλλά πάρα πολύ εξειδικευμένη. Είναι τόσο εξειδικευμένη που ε, δεν αξίζει τελικά να καλύψει και να στα capability των διαφόρων χωρών, γιατί είναι κάτι πραγματικά πολύ ιδιαίτερο και πολύ εξειδικευμένο. Άρα, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους ε, δεν επελέγησαν αυτά τα έργα και δεν καταλήξαμε να τα αξιολογούμε ως πάρα πολύ χρήσιμα. Αυτά είχα να προσθέσω. Ευχαριστώ. Και εγώ ε, θέλω να πάρω το λόγο για να μιλήσω για τον προπολογισμό. Φυσικά και υπάρχει προπολογισμό, αλλά δεν είναι προαπαιτούμενο να υποβληθεί σε εμά ο προπολογισμό. Οι συντάκτε τη πρότασης ε, καθόρισαν το, την πρόταση και τις λεπτομέρειες και το κόστο που συνεπάγεται, αλλά δεν είναι δικό μας καθήκον να αξιολογήσουμε τον προπολογισμό. Θεωρώ και υποθέτω ότι τα κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο συμπεριέλαβαν τα διάφορα στο δικό τους αμυντικό προϋπολογισμό και υπάρχει βεβαίως πολιτική λογοδοσία από αυτού. Για το θέμα της Ιρλανδίας δεν θέλω να κάνω εικασίες για το γιατί δεν προσχώρησε η Ιρλανδία σε αυτά τα έργα. Αν δεν προσχώρησε είναι γιατί θεωρούν ότι δεν ταιριάζουν τα έργα που προτάθηκαν με τις δικές τους Ιρλανδικές επιχειρησιακές ανάγκες ή άλλες. Ίσως το επόμενο κύμα έργων που ε, έρθει να θελήσει η Ιρλανδία να υιοθετήσει και να προσχωρήσει στην υλοποίηση συγκεκριμένου έργου ή οποιαδήποτε άλλη χώρια. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορώ να προβλέψω και να διατυπώσω εικασίες για τους λόγους για τους οποίους η Ιρλανδία ή οποιοδήποτε άλλο κράτος ε, δεν ε, θέλησε να συμμετάσχει στη, σε αυτά τα έργα. Να σας πω ότι με εκπλήσει αυτό το παράδειγμα με τις στρατηγικές αερομεταφορές, ότι μόνο ένα κράτος μέλος μπορεί να ε, το κάνει αυτό. Όλα τα κράτη-μέλη αναγνωρίζουν ότι υπάρχει έλλειμμα σε αυτό το τομέα Και είναι κρίμα που δεν το στηρίζουν αυτό διάφορα κράτη-μέλη. Τώρα για το κόστος. Νομίζω ότι δεν είναι σόφρον από τακτική σκοπιάς να προσθέτουμε νούμερα σε αυτές τις προτάσεις, γιατί τότε ο κλάδος θα πει να, ε, «Α, τα κράτη είναι έτοιμα να πληρώσουν τόσα χι χρήματα, ας τους τα χρεώσουμε δηλαδή». Και σε μία από τις υποστολέ στο Ελσίνκι είχα την ευκαιρία να μιλήσω με Φιλανδούς συναδέλφους που παρουσίασαν το κουάτ τους στις Βρυξέλλες και μου είπαν ότι απαντήσαμε για τα πάντα, αλλά δεν δώσαμε αριθμητικά στοιχεία και νούμερα γιατί θα τα πάρει ο στρατιωτικός κλάδος και θα τα προβλέψει, θα προβλέψει πόσα είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε. Άρα να είμαστε σόφρονες, επιφυλακτικοί με το πόσα θέλουμε να ξοδέψουμε και να αφήσουμε χώρο, περιθώριο ελιγμών για ε, αυτό το μπραντεφέρ, για αυτό το πόκερ και τη διαπραγμάτευση με τη βιομηχανία, με τον κλάδο που μετά θέλει να ε, χρεώσει ε, σε επίπεδο εμπορικό για τα προϊόντα και τις δράσεις αυτές. Θέλω να ευχαριστήσω τους ε, εισηγητές για τις απαντήσεις, για τις παρεμβάσεις, για τις παρουσιάσεις τους. Σίγουρα θα παρακολουθούμε στενά τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί αυτή η δράση. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ολοκληρώνεται η εξέταση του σημείου 12 της ημερήσιας διάταξης. Yes, yes. So, uh, the next uh, point of... Το επόμενο σημείο στη μέση διάταξη είναι και κλεισμένο το θυρών. Μπορεί αυτό το in camera να σας ε, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα έχουμε κάμερες, αλλά το αντίθετο ισχύει. Είναι και κλεισμένο το θερόν θυρών. Θα πρέπει λοιπόν όσοι δεν έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν εδώ να αποχωρήσουν από την αίθουσα. Uh, other than members and group staff and those who are entitled to to speak on this agenda item. Uh, I have already seen some assistance of MEPs leave. Είδα ήδη και ορισμένους βοηθούς ευρωβουλευτών να αποχωρούν και ο δικός μου αυτό έκανε, έδωσε το καλό παράδειγμα. Ας ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι λοιπόν. Although I have to say, in all these in-camera meetings, uh, I can often confirm what... Παρότι συχνά σε αυτές τις συνεδριάσεις ε, κεκλεισμένων των θυρών βλέπουμε ότι διαραίουν αυτούσιες ε, στον τύπο. αλλά αν κάτι είναι απόρριτο, καλύτερο είναι να το θέτουμε σε αυτό το πλαίσιο.